Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Dear members, uh, dear... Αγαπητά μέλη, αγαπητοί ομιλητές, ε, αγαπητοί συμμετέχοντες, Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ακρόαση για τα δικονομικά δικαιώματα ύποπτων και κατηγορουμένων επιτεγμάτα και το μέλλον προστασία των ατόμων στη δικονομική διαδικασία αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ένωσης και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση σήμερα εδώ σήμερα. Έχουμε διακεκριμένους προσκεκλημένους και ομιλητές ε, σήμερα για εσάς. Κάποια διαδικαστικά πρώτα απ' όλα να σα ενημερώσω ότι παρέχεται διερμηνία σε όλε τι επίσημε γλώσσε Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση τα δανέζικα, τα λετονικά και τα κροατικά. Επίσης, έχετε υπόψη σας, ε, ιδιαίτερα οι προσκεκλημένοι, ότι η ακρόαση ε, μεταδίδεται μέσω web stream και όλες οι ομιλίες εδώ καταγράφονται. Εγγράφονται και όλες οι διαδικασίες εδώ, όλες οι μας εργασίες. Για να αφήσω το χρόνο που χρειαζόμαστε για τη συζήτηση παρακαλώ τηρήστε το χρόνο ομιλία σα. Η συζήτησή μα σήμερα θα εστιαστεί στην προστασία των ατόμων στι δικονομικέ διαδικασίε ω θεμελιώδου αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ω τρόπο ε, διατήρηση τη αμοιβή εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη και τη δημοσία εμπιστοσύνη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον Ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνη, οι πολίτε όχι μόνο πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να είναι και ε, βέβαιοι γι' αυτό όταν ασκούν το δικαίωμα ελευθερής ε, κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, σήμερα εξετάζει τρεις φακέλους η Επιτροπή μας σε αυτόν τον τομέα. Πρώτος, το σχέδιο οδηγίας για τις εγγύησεις για ανήλικα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται στις ε, στην ποινική δικονομία, μια οδηγία για τη τεκμηριωθότητα και μια οδηγία για την νομική συνδρομή και τη νομική συνδρομή στις ε, διαδικασία του εντάλματος σύλληψη. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Τάρου Σπρόκνεν που θα κάνει, ή στην κυρία Σπρόκνεν που θα κάνει μια εισαγωγή. Καλώς ορίστε στην Επιτροπή μας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα. Μου ζητήθηκε να σας ε, κάνω μια παρουσίαση με τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις του μέλλοντος όσον αφορά τις δικονομικές εγγύσεις για υπόπτους και κατηγορουμένους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσω από μια υπενθύμηση των προβλημάτων που συνήθως αντιμετωπίζουμε και που είναι η αιτία που μας οδήγησε στην υιοθέτηση των μετρών αυτών. προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν ε, τα ύποπτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, όπως βλέπετε στις διαφάνειες, πρακτικές που παρακάμπτουν το δικαίωμα στη σιωπή, οι οποίες σχετίζονται στενά με την κατάχρηση της προφυλάκησης και μεγάλα διαστήματα προφυλάκησης. Θα το γνωρίζετε ότι ο πληθυσμός της φυλακές ε, που είναι προφυλακισμένος στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες είναι μικρότερος από ό,τι στις νότιες. Νομίζω 14% στη Φιλανδία, στην Αγγλία και στην Ουαλία, αλλά περίπου 30% στη Γαλλία και 60% στην Ιταλία. Ο σημαίνει ότι όταν κάποιος κατηγορείται και γνωρίζω ότι θα προφυλακιστεί για μεγάλο διάστημα. Ε, αυτό επηρεάζει το δικαίωμα στη σιωπή ενό κατηγορουμένου. Ένα άλλο ζήτημα είναι η έλλειψη πρακτικής εγγύησης του δικαιώματος ε, νομικής συνδρομής σε, στην προκατακτική φάση. Πρακτικά, διότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα υπάρχουν αρκετά καλά πρότυπα στην νομοθεσία τους αλλά το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται τα πρότυπα αυτά στην πρακτική. Ε, παρουσιάζονται ελλείψεις στην εγγύηση πρόσβασης σε πληροφορίες για υπόπτους, πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, όπως και πληροφορίες για το τι υλικό υπάρχει στη δικογραφία. Πρόβλημα λοιπόν πρόσβαση στη δικογραφία από τους υπόπτους. Τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει όσον αφορά την νομική συνδρομή αφορούν έλλειψη διαδικασιών και δομών για έγκαιρη συνδρομή. Σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν επαρκή συστήματα αυτόματης ε, νομικής συνδρομής δεν λαμβάνει το άτομο νομική συνδρομή έγκαιρα σε ένα αστυνομικό τμήμα για παράδειγμα έχει προβλήματα επιλογής ε, δικηγόρου, υπάρχει έλλειψη μηχανισμών ε, ε, εφαρμογής και πράγματα που συχνά συναντάμε στις ερευνές μας η ποιότητα της νομικής συνδρομής που παρέχεται και που έχει επίσης να κάνει με το πώς αμείβονται οι δικηγόροι που παρέχουν τη νομική συνδρομή. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, το ζήτημα της νομικής συνδρομής. Όλοι γνωρίζουμε, πιστεύω, ότι χωρίς νομική συνδρομή ε, πολλοί, οι περισσότεροι ύποπτοι κατηγορούμενοι δεν λαμβάνουν καμία νομική συνδρομή. Το 95% των υποπτών των εναγωμένων αυτών δεν δίνονται να πληρώσουν την αμοιβή για τη νομική συνδρομή οι ίδιοι και αν δείτε το πώς ρυθμίζεται η νομική συνδρομή σε εθνικό επίπεδο οι μέθοδοι εφαρμογής είναι περίπλοκες ή ασαφείς, ε, ειδικότερα κατά το πρώτο διάστημα της ε, σύλληψης από την αστυνομία. Ανεπαρκής αμοιβή λοιπόν και φυσικά ειδικότερα τώρα σε εποχές κρίσης ε, το θέμα αυτό είναι μια από τις προτεραιότητες ε, στην ατζέντα κάθε κυβέρνησης. Οι μηχανισμοί διορισμού απειλούν την ανεξαρτησία των δικηγόρων και είπε και κινδυνό οι κυβερνήσει να καθιστούν διαθέσιμη τη νομική συνδρομή μόνο μέσω συγκεκριμένων γραφείων που πρέπει να εγγραφούν για να παράσχουν συγκεκριμένη νομική συνδρομή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό φυσικά μπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα και την αυτονομία τη νομική συνδρομή που παρέχεται. Όλα αυτά έχουν συνέπειε ε, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ενό δικηγόρου, πρόσβαση δικηγόρου και για την ποιότητα της δικηγορικής συνδρομής. Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω, εδώ βλέπετε τον οδικό χάρτη στην οθόνη από τότε που το παρουσιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου αποφασίστηκε ότι αντί να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα πλήρες μέσο που θα καλύπτει όλες τις δικονομικές εγγύσεις για τους υπόπτους ε, αποφασίστηκε να υιοθετηθεί μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για τη διαπραγμάτευση των μέτρων που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη. Όπως βλέπετε στην οθόνη και όπως γνωρίζετε όλοι, η μετάφραση και η διερμηνία και η ενημέρωση για τα δικαιώματα, τις κατηγορίες και η νομική συνδρομή που συμπεριλαμβάνει την επικοινωνία με εργοδότες και τις προξενικές αρχές. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν ε, ήδη ενταχθεί στις οδηγίες και αυτή τη στιγμή αυτό που συζητείται είναι η συζήτηση περινομικής συνδρομής. Ε, συζητούνται ειδικέ εγγύησει για υπόπτους κατηγορουμένους παιδιά και αυτό που υπήρχε στην αρχή ως οδικό χάρτης, μια πράσινη βίβλος για την προφυλάκηση. Πρώτα απ' όλα, θέλω να τονίσω το εξή. Να σας πω ειλικρινά ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξίζουν συγχαρητήρια για τα όσα έχουν επιτύχει. Διότι παρά τις επικρίσεις από τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τους δικηγόρους σε όλα τα επίπεδα, λέγοντας ότι είναι αδύναμα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν λόγω των διαπραγματεύσεων, παρόλα αυτά έχουν επιτευχθεί πολλά, αν σκεφτεί κανείς πώς είχε καταστήσει το 2007 όπου η απόφαση πλαίσιο για τις δικονομικές εγγύησεις ε, ήταν εντελώς αδρανής, ε, δεν εξέταζε κανένας. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν πρώτα απ' όλα, πραγματοποιήσαμε μελέτη που ονομάζεται Inside Police Custody με το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ και άλλους εταίρους για να εξετάσουμε την πρακτική αποτελεσματικότητα μέτρων σαν αυτά, όπω μετάφραση και διερμηνία, δικαίωμα στην ενημέρωση, δικαίωμα στην νομική συνδρομή και δικαίωμα στη σιωπή σε τέσσερι χώρε. κάτω χώρε: Γαλλία, Αγγλία και Ουαλία. Δεν μπορεί να πούμε ξεχωριστή χώρα βέβαια και στη Σκωτία που έχει όμω ξεχωριστό δικαστικό σύστημα από την Αγγλία και η Ουαλία. Ε, πρόκειται για μια εμπειρική μελέτη Βάλαμε ανθρώπους σε αστυνομικά τμήματα, ερευνητές για αστήματα 5-6 μηνών που εξέταζαν τι ακριβώς γίνεται στην πρακτική και πώς ακριβώς ε, διαφυλάζονται αυτά τα δικαιώματα στην πρακτική και τι είδους προβλήματα προέκυπταν με αυτά τα δικαιώματα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε Ε, σε μια εποχή όπου η περίοδη υλοποίηση των οδηγιών που μόλις είχαν υιοθετηθεί δεν είχε ακόμα λήξει, οπότε ήταν μια έρευνα που λάμβανε χώρα σε φάση που δεν είχαν ακόμα υλοποιηθεί οι οδηγίες αυτές. Να σας παρουσιάσω κάποια σημαντικά στοιχεία που ανακαλύψαμε και που ελπίζουμε να έχουν βελτιώσει οι οδηγίες. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη μεταφράση και τη διερμηνία. Πρακτικά, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει κάποια διαδικασία αξιολόγηση της ανάγκης ύπαρξη μεταφράσης και Και η οδηγία βελτίωσε τα πράγματα. Υπάρχει διορθωτικό μέτρο διαθέσιμο σε περίπτωση όπου ένα ύποπτο χρειάζεται μετάφραση εγγράφων και δεν χορηγείται αυτή η μετάφραση. Όσον αφορά το δικαίωμα στην ενημέρωση, αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι στι περισσότερε περιπτώσει η ενημέρωση περί δικαιωμάτων παρέχεται στους υπόπτους αλλά σε μια χρονική στιγμή και με τέτοιο τρόπο που οι ύποπτοι που είχαν συλληφθεί στο αστυνομικό τμήμα δεν προλάβαιναν να σκεφτούν και να αποφασίσουν τι δυνατότητες είχαν, τι δυνατότητες προσφέρονταν ε, μέσω αυτής της ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να έχουμε στο νου μας στο πλαίσιο των οδηγιών αυτών, ειδικότερα για την οδηγία περί δικαιωμάτων ενημέρωσης ε, και κατά την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά το δικαίωμα στην νομική βοήθεια και νομική συνδρομή, εξετάσαμε περιπτώσεις όπου η νομική συνδρομή ήταν δυνατή κατά την ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα και, τις, και υπήρξε ένα σύστημα που εφαρμόζεται στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία και σε ένα σύστημα όπου δεν υπήρχε δυνατότητα να είναι παρόν δικηγόρος κατά την ανάκριση. Πράγμα που ακόμη συμβαίνει στις κατοχώρε. Το ανώτατο δικαστήριο στις κατοχώρες δεν θέλει να λαβεί καμία απόφαση για αυτό το θέμα πριν ενσωματωθεί η οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Τι φοβόμαστε Πρέπει να το ξέρετε. Όταν υπάρχει δικηγόρος παρόν κατά την ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα, ε, μπορεί τότε ο ύποπτο να επικαλεστεί το δικαίωμά του στη σιωπή. Η αστυνομία στη Γαλλία, στις κατοχώρες αλλά και στο Βέλγιο το φοβούνται αυτό. Γιατί παρατηρήσαμε ότι το 50 έως 60% των υπόπτων παρετούνται του δικαιώματος στη ΣΥΟΠΗ... δίνουν πληροφορίες στην αστυνομία ακόμα και αν έχουν ενημερωθεί πολύ καλά για το τι, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει παρόν δικηγόρος και παρόλα αυτά πολλοί υπόπτοι παρετούνται του δικαιώματος στην νομική συνδρομή διότι πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους και δεν θέλουν να αποσχοληθεί κάποιο δικηγόρος. Το ίδιο ισχύει για το δικαίωμα στη ΣΥΟΠΗ. Ελάχιστα είναι τα αποτελέσματα που βλέπουμε όσον αφορά τα ποσοστά απαραίτησης ε, του δικαίωματος ε, στη σιωπή. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένας δικηγόρος, ακόμη και ένας δικηγόρος είναι παρόν, ε, οι υποπτοί δεν συνεργάζονται με την αστυνομία πλέον, αλλά όταν συνεργάζονται, η απόφαση που λαμβάνουν βγαίνεται βάσει πιο καλή ενημέρωσή τους. Να σας δείξω τώρα τι βλέπουμε για το μέλλον διότι αυτά που συζητάμε είναι εγγύσεις για τα παιδιά, το τεκμήριο αθότητας και νομική συνδρομή. Αυτό που θέλω να δηλώσω εδώ ως ανησυχία είναι ότι γενικά έχουμε διάφορες ε, πιθανές δυσκολίες σε αυτή τη βηματική προσέγγιση για το μέλλον. Αυτό έχει να κάνει με την συνοχή μεταξύ των οδηγιών. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα μικρά δικήματα τις περιπτώσεις μη εφαρμογή των οδηγιών. Αυτό πραγματικά αποτελεί πρόβλημα. Διότι, ο ορισμός του μικρού αδικήματος είναι αρκετά σαφής. Δεν υπάρχει στις αιτιολογικές σκέψεις. Παραμένει σαφής και στα άρθρα. και στο πλαίσιο της οδηγίας που αφορά την πρόσβαση σε δικηγόρο εκεί έγινε μεγάλες συζητήσεις για το κατά πόσο πρέπει να εμπλακεί η δικηγόρο σε όλες τις περιπτώσεις όπως περίπτωση διακίνησης ή σε μικρά αδικήματα. Ε, συμφωνήθηκε λοιπόν εκεί ότι η σε μικρα δικηματα ελευθερίας είναι πραγματικά μια κατάσταση όπου πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παροχής συμβουλών από έναν δικηγόρο. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση των μικρών αδικημάτων ξεκινά και πάλι ε, στο πλαίσιο της οδηγίας ε, ε, περιεγγύσεων για τα παιδιά. Και το ερώτημα εκεί είναι κατά πόσο εδώ τα πράγματα πρέπει να διαφέρουν από τη γενικότερη οδηγία πρόσβαση σε δικηγόρο, κατά πόσο οι εγγύσει πρέπει να είναι διαφορετικέ για τα παιδιά. Και εδώ επαναρχόμαστε στο ζήτημα τη ασυνοχή μεταξύ των οδηγιών. Επίση, η χρήση τη επίσημη νομική ορολογία είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιληφθούμε. Λέξει, όπω σύλληψη, ύποπτο, εναγόμενο, μπορεί να σημαίνουν διαφορετικά πράγματα σε κάθε δικαιοδοσία και αν αυτό σχετίζεται με πότε εφαρμόζεται η οδηγία υπάρχει περίπτωση να εφαρμόζεται σε διαφορετική στιγμή σε ένα κράτος μέλος και σε διαφορετική στιγμή σε ένα άλλο κράτος μέλος. Πιστεύω λοιπόν ότι σκόπιμο θα ήταν να επιλέγουμε γλώσσα στην οδηγία που να είναι πολύ ρεαλιστική, να βασίζεται σε γεγονότα συγκεκριμένα και όχι να βασίζουμε την ερμηνεία της οδηγίας για να ορίσουμε τη στιγμή στην οποία ε, μπορεί να αρχίσει να ισχύει ένα δικαίωμα που προβλέπεται στην οδηγία. Τρίτον, ε, άλλη μια γενική δυσκολία είναι ο ορισμός του πεδίου εφαρμογή ε, της οδηγίας. Για παράδειγμα, έχουμε διαφορετική γλώσσα στην οδηγία νομικής συνδρομής η οδηγία ισχύει από τη στιγμή που γνωρίζει ο ύποπτος από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μέσω επίσημης ειδοποίησης με άλλο τρόπο ότι είναι ύποπτος ή κατηγορείται ε, για τη διάπραξη ενός ποινικού αδικήματος. Αυτή είναι μια ευρεία ε, αλλά ρεαλιστική ε, περιγραφή αλλά στην οδηγία για το τεκμήριο αθότητας λέει ότι η οδηγία εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται στο πλαίσιο ποινική δικονομία. Κάτι πολύ πιο ασαφέ ε, όσον αφορά τον ορισμό του πεδίου εφαρμογή. Και μετά φυσικά έχουμε τι εξαιρέσει. Σημαντικό κομμάτι. Και έχω δει ότι τώρα προτείνεται νομοθεσία για τα δικαιώματα πρόσβαση σε δικηγορο στις και εκεί έχω δει ήδη ότι στην νομοθεσία οι εξαιρέσει που υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία έχουν οριστεί με ευρύ τρόπο, με πιο ευρύ τρόπο από ό,τι αναφέρεται στην οδηγία. Για να σας δώσω μερικά παραδείγματα, η οδηγία για το δικαίωμα προσβάση σε δικηγόρο έχει κάποια καλά στοιχεία ότι το πεδίο εφαρμογή είναι ανεξάρτητο από τι θέσει ελευθερία και ότι ισχύει πριν και κατά τη διάρκεια όλων των ανακρίσεων. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά και θα κάνει μεγάλη διαφορά σε πολλά κράτη-μέλη. Οι προβληματικέ πτυχέ είναι τι σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή δικηγόρου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. στι κάτω γίνεται η συζήτηση για το πότε παρεμβαίνει ο δικηγόρος που κάθεται, αν κάθεται δίπλα στον ε, ύποπτο, αν μπορεί να έχει επαφή με τα μάτια και τα λοιπά. Και μετά και το θέμα των εξαιρέσεων αποτελεί πρόβλημα, αλλά το ανέφερα ήδη και μετά. Μια άλλη σημαντική πτυχή πιστεύω είναι ο συσχετισμός των δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, όλες αυτές οι οδηγίες συσχετίζονται μεταξύ τους. Ε, αν δει κανείς το δικαίωμα για ενημέρωση και τη στιγμή παρέχεται ενημέρωση σε έναν ύποπτο, ε, όλα αυτά ε, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αν ο ύποπτος θα παραιτηθεί ή όχι του δικαιώματος σε δικηγόρο. Η στιγμή λοιπόν που παρέχεται η ημερομηνία πρέπει να είναι τέτοια ώστε μετά να έχει κάποιο χρόνο ο ύποπτος να δει αν θέλει δικηγόρο ή όχι στο Βέλγιο δεν μπορεί να παραιτηθεί τέτοιου δικαιώματο ο ύποπτο αν δεν έχει μιλήσει πρώτα με δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι του χρειάζεται κάποιο χρόνο. Να του δοθούν οι πληροφορίε, να γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, να σκεφτεί κατά πόσο θέλει να παραιτηθεί του δικαιώματο και αυτό είναι εντελώ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία και στην Ουαλία. Εκεί του ρωτούν θέλετε δικηγόρο και αν ο ύποπτο πει όχι, του λένε τότε γιατί όχι και αν ο ύποπτο πει δεν με νοιάζει, θα τα καταφέρω μόνο μου, τελείωσε η υπόθεση. Δεν υπάρχει δηλαδή χρόνος μεταξύ της παράδοσης πληροφορίας και της παρέτησης από το δικαίωμα. Μετά η πρόσβαση, το δικαίωμα πρόσβαση στη δικογραφία. Και αυτό σχετίζεται με το τι μπορεί, πώς μπορεί να βοηθήσει ένας δικηγόρος ο, συμβουλεύοντας τον πελάτη του και για το κατά πόσο πρέπει να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο υποπτός τι είδους πληροφορίες έχει στην κατοχή της αστυνομία. Και αυτό είναι κάτι νομίζω που ρυθμίζεται με, ε, στο πλαίσιο της πρόσβασης στη δικογραφία, στην οδηγία περί ενημέρωσης και σχετίζεται με τη δυνατότητα ε, λήψης δικηγορικής ε, υποστήριξης. Θέλω να σα προσθέσω κάποια ερωτήματα που θα οδηγήσουν σε συζητήσει όσον αφορά την πρόταση για μια οδηγία για τι δικονομικέ εγγυήσει για παιδιά. Αυτό που είναι σημαντικό να συζητήσουμε είναι η νομική συνδρομή για τα μικρά αδικήματα. Γιατί θα μπορούσε κανεί να σκεφτεί ότι όταν έχουμε παιδιά ω υπόψη, αλλά αυτό βέβαια ισχύει και για ενήλικε, νοούνται διαφορετικά τα μικρά αδικήματα περιλαμβάνονται στα ποινικά μητρώα. Τι σημαίνει για το μέλλον ενός παιδιού μια τέτοια κατηγορία. Όταν θα χρειαστεί να βρει μια δουλειά για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει μια τελείως διαφορετική πτυχή που επηρεάζεται από τον ορισμό των μικρών αδικημάτων. Και επίση ε, ρωτήσαμε γιατί να γίνονται εξαιρέσει ε, για την ηχητική ή οπτική εγγραφή τη ανάκριση από την αστυνομία για τα μικρά δικήματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνονται τέτοιε εξαιρέσει. Όσον αφορά την οδηγία για το τεκμήριο αθωότητας, ε, είναι προβληματική η διάκριση μεταξύ ποινική και διοικητική διαδικασία και κυρώσεων που βρίσκεται στην αιτιολογική σκέψη 6. Γιατί αυτό που βλέπουμε σε πολλέ χώρε είναι ότι Υπάρχει μια μια μεταφορά από την ε, ποινική προς τη διοικητική διαδικασία και μπορεί να υπάρχουν σημαντικές κυρώσεις στη διοικητική ε, διαδικασία. Γιατί να κάνουμε λοιπόν τέτοια διάκριση. Και μετά τι γίνεται σε σχέση με τη θέση ενός μάρτυρα ή ενός συγγενούς όσον αφορά το προνόμιο ε, που έχει κάποιο να μην ε, ε, υπάρξει μάρτυρα. Μετά έχουμε την οδηγία για την νομική συνδρομή. Αυτή θα αποτελέσει το θεμελιώδη λίθο για την αποτελεσματικότητα και των υπολείπων οδηγιών. Η έννοια της προσωρινής νομικής συνδρομής πιστεύω είναι πολύ καλή ιδέα για να δώσει μια λύση στις περιπτώσεις που πραγματικά απαιτείται νομική συνδρομή κατά την πρώτη φάση μιας αστυνομική έρευνας όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κάποια μεγάλη διαδικασία αξιολόγηση του κατά πόσο ένα άτομο πρέπει να έχει νομική συνδρομή. Και φυσικά μετά υπάρχει και ο περιορισμό τη τέρηση τη ελευθερία και αυτό εξαρτάται. Πρέπει να το συζητήσετε σε σχέση με τα μικρά αδικήματα. Και έχει να κάνει με τον ορισμό του μικρού αδικήματο. Το συμπέρασμά μου λοιπόν έχει ω εξή ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επικοδομητική πραγματικά, αλλά ο διάλογος είναι στις λεπτομέρειες. Και προκύπτουν νέα ερωτήματα. Αυτό είναι το τελευταίο που έχω να πω. Πώς αυτές οι οδηγίες για τις δικονομικές εγγύσεις επηρεάζουν τις οδηγίες που βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση. Πώς επηρεάζεται η διασυνοριακή συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων πώς επηρεάζει το δικαίωμα σε νομική συνδρομή και δικαιή δίκη γενικότερα και πώς σχετίζονται όλα αυτά με τη νομική συνδρομή το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας πώς σχετίζεται με τη νομική συνδρομή όταν συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία σε μια άλλη χώρα σε σχέση με τη νομική συνδρομή. Αυτά ήθελα να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. ευχαριστούμε πολύ κυρία Σπρόγκεν. Θα σας έκοβα βέβαια όπου να είναι γιατί είχατε ξεπεράσει αρκετά τον ε, χρόνο. Αλλά ήταν ενδιαφέρον το κομμάτι κοινό της ομιλίας σας για την παρέμβαση από απεξένωση και δεν ήθελα να σας διακόψω. Θα ζητήσω τώρα από τους ε, εισηγητές να πάρουν το λόγο και να προεδρεύσει ο ένας μετά τον άλλον των σχετικών συνεδριών. Έχω συναδέλφους ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Westminster. Σηκώστε τα χέρια σας να σας δούμε χθες ε, δεν ήταν τόσο ειρηνική η ατμόσφαιρα όταν συζητούσαμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, Σύλληψης. Δεν είναι τόσο ήρεμα πάντα τα πράγματα. Έχουμε ακαδημαϊκούς ε, και δικηγόρους σήμερα. Γι' αυτό είναι πιο <coughs> ήσυχα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σπρόγκεν για την πολύ διαφωτιστική αυτή εισαγωγή και τώρα θα ζητήσω από τους συζητητές μας για τα τρία θέματα να έρθουν στο βήμα. Πρώτα απ' όλα την ε, Κατρίνα και κύριοι Πικάλ και Πατανέ. As, um, Katerina is Μέχρι να έρθει η Κατρίνα Τσινίκη να πω ότι είναι η συγγήτρια για την οδηγία για τα παιδιά. E Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, κύριε Μωράης και βέβαια θέλω να καλωσορίσω και όλους τους προσκεκλημένους και συνοδέλφους. Νομίζω ότι σήμερα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχουμε μια πολύ καλή δυνατότητα για να εμβαθύνουμε σε κάποια ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας αλλά και για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου εν γέννη. Είχαμε πει στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής ε, Λίμπε στις 16 Οκτωβρίου ότι η πρόταση οδηγίας για τους ανηλίκους ε, που είναι υποπτικά κατηγορούνται εντάσσεται σε μια δέσμη μέτρων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων. υπόπτων ή κατηγορουμένων. Στο τομέα της ποινικής δικονομίας. Στις 15 Φεβρουαρίου του 2011 είχαν εγκριθεί και κάποιες διατάξεις σε σχέση με, τα, με τους ανηλίκους. Υπάρχουν διατάξεις που έχουν εγκριθεί, κάποιες είναι υποσυζήτηση ακόμα. Μιλάμε για μέτρα που έχουν όλα την ίδια νομική βάση και τον ίδιο στόχο, δηλαδή να έχουμε κάποιες ελάχιστες διατάξεις που θα ισχύουν για όλους όσους είναι υποπτή κατηγορούνται στο πλαίσιο Οικονομικών διαδικασιών. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Και βέβαια τα κράτη-μέλη μπορούν, αν θέλουν, να εισαγάγουν διατάξεις που να ενισχύουν την προστασία των ατόμων αυτών. Σε ό,τι αφορά την οδηγία, για την οποία είμαι συγγήτρια, οδηγία για τους ανηλίκους, θα την ε, αποκαλώ για χάρη συντομίας, θέλουμε να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Πρέπει να υπάρχουν διάφορες ασφαλιστικές δικλείδε. Το δικαίωμα ενό ανηλίκου σε δίκαιη δίκη δεν είναι όμω εγγυημένο επαρκώ σήμερα ή τέλο πάντων όχι με τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν μια έλλειψη που πρέπει να διορθωθεί. Εξού και η οδηγία αυτή για τους ανηλίκους περιλαμβάνει σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες. συντομία θα τις αναφέρω. Δικαίωμα ενημέρωσης και για τον ανήλικο, αλλά και για οποιονδήποτε ενήλικο είναι, έχει την επιμέλεια την κυδαιμονία του ανηλίκου. Δεν μπορεί ε, να υποκαταστήσει αυτό το δικαίωμα το δικαίωμα σε ένα δικηγόρο υπεράσπισης. Επίσης υπάρχουν και άλλα δικαιώματα, ετικών εξτάσεων κτλ. Σε ό,τι αφορά τη στέρηση ελευθερία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρό το χρονικό διάστημα. Και πολλές άλλες ασφαλιστικές δικλείδες. Ίσως και με τις τροπολογίες μας θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις σχετικές διατάξεις. Και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να μάθουμε πολλά για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, ακούγοντας τις απόψεις και τις ε, παρεμβάσεις ειδικών από τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα που σίγουρα θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες Έχουμε μαζί μας τον Δ. Ντανιέλ Πικάλα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης ε, δικαστικών για ανηλίκους και οικογένειες. Τον ευχαριστώ που βρίσκεται εδώ στην ακρόαση της Επιτροπής μας. Ο Δ. Πικάλ από την εμπειρία του ως δικαστής για ανηλίκους έχει αντιμετωπίσει υποθέσεις σαν αυτές που αποτελούν το αντικείμενο της οδηγίας μας. Ε, συνεπώς η παρέμβασή του θα είναι πολύ σημαντική για μας και του δίνω το λόγο και τον παρακαλώ βέβαια να περιοριστεί στα όρια των 10 λεπτών ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιαγράμμα των εργασιών μας. Ε, παρακαλώ κύριε Πικάλ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τα δεκάλεπτα λεπτά και έχω να πω πολλά. Θα προσπαθήσω να είμαι πάντως συνοπτικός. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης ε, Δικαστών και Επιμελητών ε, Ανηλίκων ε, του οποίου, της οποίας προεδρεύω. Έχουμε κάνει ήδη πολλή δουλειά η οδηγία έχει να κάνει και με, το, ε, με την εκπαίδευση των ε, δικαστών ανηλίκων και των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Αφήνει όμως εκτός το θέμα της δημιουργίας κάποιων ε, δικαστηρίων για ανηλίκους και για την κατάρτιση δικαστών που θα ασχολούνται ειδικά με τα θέματα των ανηλίκων. Αυτό δεν μας ικανοποιεί. Κάτι άλλο που δεν μας ικανοποιεί είναι ότι η μελλοντική οδηγία δεν μιλάει για την ελάχιστη ηλικία ποινική ευθύνη, αλλά σε ό,τι αφορά την εφαρμοσιμότητα της οδηγίας υπάρχει ένα μέγιστο όριο ηλικία. Οπότε και θεωρείται ενήλικος πλέον. Είναι δηλαδή κάπως πιο αφηρημένη η έννοια του ανηλίκου. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή τώρα του σχέδιου οδηγίας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ασάφεια στην αρχή στο κείμενο σε ό,τι αφορά το όριο ηλικίας εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Στα άρθρα 2 και 3 προστίθεται μία φράση ότι κάθε πράξη που διαπράτεται από ένα παιδί πριν φτάσει στην ηλικία των 18 ετών πρέπει να επιτρέπει να διευκρινιστεί αυτή η κατάσταση κατά την άποψή μας. Γιατί μιλάει το κείμενο από τη στιγμή που είναι ύποπτο ή κατηγορείται ένα παιδί ή από τη στιγμή που ενημερώνεται για ότι είναι ύποπτο ή κατηγορείται. Τότε αρχίζει να ισχύει οδηγία και βέβαια αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε το παιδί που έχει διαπράξει το αδίκημα μπορεί να έχει μέχρι ότου επιβεβαιωθούν τα πραγματικά περιστατικά να έχει ενηλικιωθεί. Το θέμα είναι η στιγμή διάπραξη του αδικήματος. Τι ηλικία είχε τότε το παιδί και από εκεί ξεκινά και η οδηγία να ισχύει. Αν υπάρξουν αυτές οι διευκρινήσεις, νομίζω ότι θα είναι πιο σαφές το παιδί εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Και αν το παιδί είναι λιγότερο από 18, όταν διέπραξε το αδίκημα, τότε βέβαια θα πρέπει να ισχύει γι' αυτό η οδηγία. Μέχρι το τέλος της διαδικασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του σχεδίου που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ιδίως οδηγίες του Συμβουλίου, για την μη εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Άρθρο 6 λέει η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες που αφορούν παιδιά που έχουν ε, διαπράξει ένα αδίκημα, μια παράβαση, όταν θα μπορούσε να μην επιβληθεί ποινική ε, κύρωση, αλλά περιοριστικά μέτρα κατά του παιδιού. Και υπάρχει ε, ο όρος μπορεί, μπορούν. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή κατά πόσο θα υπάρξει ποινική κύρωση ή όχι. Η γαλλική νομοθεσία για παράδειγμα, <clears throat> σε ό,τι αφορά τους νεαρούς ανήλικους παραβάτες έχει κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις και στον τελικό βαθμό μπορεί να υπάρξει ποινική κύρωση για τον ανήλικο, αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε όταν ξεκινάει δίκη. Γιατί στην αρχή ο δικαστής θα προσπαθήσει να βρει ε, μία λύση παιδευτική. Αν δεν καταλήξει λοιπόν ε, με ποινική κύρωση η διαδικασία δεν μπορούμε να ε, προσφύγουμε στην οδηγία. Και ποια είναι αυτά, ποια είναι αυτοί οι περιορισμοί. Μιλάμε για μέτρα που μπορούν να δικαιώσουν μέχρι και σε στέρηση ελευθερία, σε ένα ίδρυμα δηλαδή να μπει το παιδί. Φυσικά και δεν μπορούμε να έχουμε διαδικαστικές εγγύησεις ε, στην περίπτωση αυτή. Η Βελγική νομοθεσία, παράδειγμα, προβλέπει σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους μέχρι 16 ετών δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων. Τα παιδευτικά μέτρα, σοφρονιστικά μέτρα μόνο επιτρέπονται, αλλά υπάρχει δυνατότητα να εγκλειστεί σε ένα κέντρο στερητικό ελευθερίας. Άρα δεν εφαρμόζεται η οδηγία εκεί αφού δεν πρόκειται για ποινική κύρωση. Κριτήριο δεν θα έπρεπε να είναι η στέρηση ελευθερίας λοιπόν. Γιατί έτσι γίνεται αυτή η διάκριση και καταλαβαίνουμε κατά πόσο πρέπει να εφαρμόσουμε τα ηχέγγυα αυτά τις εγγύσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ε, να έχει συνδρομή δικηγόρου, άρθρο 6 το παιδί, φυσικά και υπάρχει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, θα πρέπει να έχουν ένα νομικό παραστάτη τα παιδιά, αλλά υπάρχει και το 6α που λέει ότι σε περιπτώσεις που γίνονται ανακρίσεις από τις αστυνομικές αρχές ή από μια κατασταλτική αρχή, ναι, αλλά εκτός αν είναι δυσανάλογο και αναφέρει κάποια στοιχεία μετά αυτό το άρθρο. Πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ε, η βαρύτητα του αδικήματος, ε, η μέγιστη ποινή. Άρα υπάρχουν, υπάρχει αοριστία Υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από την αρχή τη διαδικασία. Δεν είναι όμω αυτό δυνατό από την αρχή μια δίκη πάντα. Μπορεί μια δίκη αρχικά να μην φαίνεται πολύπλοκη, αλλά να προκύψουν άλλα στοιχεία στη διάρκεια τη ε, ανακριτική διαδικασία και να γίνει πολύπλοκη δίκη. Όμω έτσι θα μπορούσε να έχει στερηθεί τη παρουσία δικηγόρου το παιδί. Υπάρχει και ένα β' μικρό, λέει όταν ε, στερούνται ελευθερία, εκτό αν θεωρείται... ότι θα είναι σύντομη διάρκεια η στέρηση ελευθερία. Τι θα πει όταν υποτίθεται ότι θα είναι σύντομη διάρκεια. Και αυτό είναι προσέγγιση. Μπορεί να υποθέτουμε ότι στην αρχή θα είναι σύντομη διάρκεια, αλλά τι θα πει αυτό, κάποιε ώρε, κάποιε μέρε, κάποιε εβδομάδε. Και εδώ δεν είναι σαφή η διάρκεια. Υπάρχει μια οριστία. Ατυχή. Η παρουσία δικηγόρου θα ήθελα να πω ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα η απόφαση κατά της Τουρκίας 27 2008 λέει ότι δεν είναι μία πρόσβαση στο δικαίωμα, πρέπει να είναι πραγματική η παρουσία. Τώρα, αυτά τα μικρά δικήματα, πτέσματα, όπως παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κτλ. Ε, δεν πρέπει να είμαστε εδώ λίγο λογικοί τι κριτήρια χρησιμοποιούμε. Και πρέπει να πω ότι η Γερμανία, σε ένα σημείο που με έχει διαβιβάσει λέει ότι το 70% των ποινικών διαδικασιών ανηλίκων ε, καταλήγουν χωρίς επίσημη τιμιγορία, χωρίς επίσημη απόφαση. Γιατί είναι κάπως τετριμένες οι υποθέσεις. Και από δικαιοδοτικές πλευράς, τα δικαιώματα πρέπει να επιβεβαιώνονται δεν υπάρχουν ε, πολύ πιο μεγάλες λεπτομέρειες για τους ανηλίκους, ισχύουν ότι ε, όσα ισχύουν για τους ενηλίκους κυρίως. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 7, 8 και 9, πράγματι πρέπει να γίνει ε, η εξέταση προσωπικότητας από επαγγελματίες. χωρίς να ξεκινήσουν ιατρικές διαδικασίες, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο όμως. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, βέβαια και άλλες χώρες έχουν κάποιες εκπαιδευτικές, κοινωνικο-εκπαιδευτικές υπηρεσίες που είναι εξειδικευμένες και μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή. Ιατρική εξέταση, ιατρική εξέταση από γιατρό. Αυτό πρέπει να προβλέπετε, έτσι προβλέπει η Κομισιόν τουλάχιστον, αλλά είναι πιο περιοριστικό το Συμβούλιο και αναφέρει κάποιες περιπτώσεις όπου αυτό δεν θα ήταν αναγκαίο. Θα έπρεπε να αποδειχθεί όμως ότι η ψυχική, η σωματική υγεία του παιδιού δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Πώ θα ξέρουμε αν δικαιολογείται ή όχι, δεν πρέπει να προηγηθεί μια ιατρική εξέταση. Γίνεται πλήρη αναστροφή του βάρου απόδειξη. Φυσικά και πρέπει να προηγηθεί η ιατρική εξέταση για να διαπιστωθεί αν το παιδί είναι σε καλή ψυχική σωματική κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάκριση, Υπάρχει αυτή η οπτικοακουστική ηχο... Ε, καταγραφή, ηχογράφηση λοιπόν ε, και μαγνητοσκόπηση της ανάκρισης. Η Γερμανία ήθελε πιο πολύ ε, να γίνουν σεβαστά δικαιώματα των ανηλίκων. Βλέπω ότι τρέχει ο χρόνος, άρα κατά λίγο σύντομα, σε ό,τι αφορά την ειδική μεταχείριση για την κράτηση, την προφυλάκηση. Η οι συνθήκες κράτησης δεν αναφέρονται διαμακρών στο σχέδιο οδηγία. Το άρθρο 12 προβλέπει διαχωρισμό ενηλίκων-ανηλίκων. Αλλά υπάρχουν ε, και κάποιες, ε, κάποια παραθυράκια εδώ. Δεν έχω άλλο χρόνο, βλέπω στη διάθεσή μου. Είχα κι άλλα να πω, Φαντάζομαι θα μπορούσα να τα προσθέσω μετά από τι ερωτήσει που θα μου υποβληθούν. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Πικάλα για τις πολύ ενημερωτικές του παρατηρήσεις. Στο πλαίσιο της συζήτησης ε, θα έχετε δυνατότητα να εμβαθύνετε και περισσότερα. Δίνω τώρα τον λόγο στην καθηγητρία κυρία Βάνια Πατανέ που διδάσκει δικονομικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια και ειδικεύεται στο δίκαιο για ανελίκους. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς για αυτή την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω με μία σκέψη. Κάθε εγγύηση αντιστοιχεί σε έναν περιορισμό στην άσκηση μιας εξουσίας και όταν ρυθμίζεται πρέπει να ρυθμίζεται βάσει της αξίας που υποτίθεται ότι προστατεύει. Στον τομέα της, ε, του ποινικού δικαίου αφορά τη θυσία που υποτίθεται ότι πρέπει να επιβάλλουμε σε ένα μηχανισμό όπως η ποινική δικονομία για την προστασία κάποιων πρωταρχικών απαιτήσεων. οι τεχνικές επιβεβαίωσης ενός εγκλήματος δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τα θεμελιώδη δικαιώματα ενός ατόμου. Δεδομένης αυτής της σκέψης θα ήθελα να υπογράψω τώρα μια θεμελιώδη πτυχή που σε κάποιο βαθμό συζητείται όταν αναλύουμε τα προβληματικά σημεία της πρότασης οδηγίας. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, εμείς δεν έχουμε δίκτες που να μας λένε ακριβώς ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας δίκαιης δίκης ανηλίκου. Η αναφορά που γίνεται στις εγγύσεις για περί δίκαιης δίκης είναι αυτή που περιλαμβάνεται στους ε, ευρωπαϊκούς χάρτες και σε πολλούς ε, χάρτες θεμελιδών δικαιωμάτων των εθνικών νομοθεσιών, αλλά δεν έχουμε ακριβή ιδέα του τι σημαίνει δίκαιη δίκη ανηλίκου. Γι' αυτό τον λόγο, με αυτή την ιδέα της δίκης δίκης για ανηλίκους, είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι πρέπει να συνδέεται πάντα με έναν θεμελιώδη παράγοντα ότι η ποινική δίκη ακόμα και όταν δικάζεται ένας ανηλικός δεν πρέπει να χάνει τα χαρακτηριστικά του ως μέσου επιβεβαίωσης ποινικών αδικημάτων. Ας προσέξουμε η ποινική δικονομία για τους ανηλίκους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μια ευκαιρία για παρέμβαση κοινωνικο-παιδαγωγική στο, προς το ανήλικο. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη πνευματική διαδικασία, διαδρομή για την νομική επιβεβαίωση γεγονότων και ευθυνών. Συνεπώς η τήρηση των κανόνων της δίκαιης δίκης και στον τομέα των ανηλίκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να διασφαλίζεται η το δίκαιο της απόφασης. Επειδή κάθε εξαίρεση συνεπάγεται απαραίτητα μείωση των εγγυήσεων, αν να δούμε τις επιμέρους εγγυήσεις που αναφέρονται στην οδηγία, πρέπει να γνωρίζουμε σαφώς στο νου μας ποιος είναι ο σκοπός της εγγύησης ώστε στη συνέχεια να μπορούμε με κάποιο τρόπο να ισορροπήσουμε, να προσαρμόσουμε την εξαίρεση. Είναι πολύ επικίνδυνο παρότι αναπόφευκτο να συνδέσουμε τις εξαιρέσεις με πολύ ασαφείς έννοιες που δεν έχουν καθοριστεί επακριβώς. Ξεκινώντας από την έννοια της προστασίας των συμφερόντων του ανηλίκου που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά σε αυτή την πρόταση οδηγίας όπως και σε πολλά έγγραφα διεθνή η έννοια των συμφερόντων του ανηλίκου είναι κάτι πολύ ευρύ. Δεν μπορούμε να το ορίσουμε επακριβώς, αλλά εκχωρείς τον δικαστή μία ε, ε, διακριτική ευχέρεια τεράστια. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν οι εξαιρέσει να μην αιτιολογούνται μόνο από μια γενική αναφορά στα συμφέροντα του ανηλίκου, ας έχουμε στο νου μας το σκοπό, τον απότερο σκοπό της εξαίρεσης, ώστε να προσαρμόζουμε την εμβελία της ανάλογα. Ας περάσουμε τώρα στο να εξετάσουμε κάποια πιστεύω εγώ σημαντικά στοιχεία των επιλεγών που έχουν γίνει μέσω αυτής της πρώτης οδηγίας που ούτως ή άλλως έχει κάποιες προβληματικές πτυχές. Πρώτα απ' όλα το πεδίο εφαρμογή της ε, οδηγίας. Το άρθρο 2 λέει ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με μέτρα προστασίας ή μέτρα εκπαίδευσης δεν θα εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας και έτσι η οδηγία αυτή περιορίζεται σε άτομα που ανακρίνονται, σε ύποπτα ή που είναι κατηγορούμενοι στο πλαίσιο μιας ποινική διαδικασίας. Δηλαδή εδώ εξαιρούνται τα μικρά αδικήματα που δεν εξετάζονται από έναν ποινικό λόγο ή περιπτώσεις όπου ένας ανηλίκος έχει διαπράξει κάτι που είναι αδίκημα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αλλά που δεν ε, οδηγεί σε διαδικασίες που μπορεί να καταλήξουν σε κάποια ποινική κύρωση, αλλά που μπορούν να συνεπάγονται την επιβολή περιοριστικών μέτρων, όπως μέτρα προστασίας, διορθωτικά, παιδευτικά μέτρα, για την πρόθεση της ε, ε, βελτίωσης της συμπεριφοράς του ανηλίκου. Εδώ θέλω να σε πιστήσω την προσοχή ότι υπάρχει ο κίνδυνος όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά αυτή η υποβάθμιση του παρέμβαση μπορεί να θεωρηθεί ως νομιμοποίηση της μείωσης του επίπεδου εγγύσεων. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Εμείς όταν μιλάμε για ανηλίκους πρέπει να έχουμε στο νου μας ένα μη τυπικό ουσιαστικό προφίλ, μια μη τυπική ουσιαστική εικόνα της προστασίας και συνεπώς της αιτιολογίας που μπορεί να οδηγήσει στην εξαίρεση. Ανεξάρτητα λοιπόν από την υπόθεση όπου εφαρμόζεται η στέρηση της ελευθερίας, και από την ετικέτα που επικολλάται σε ένα τέτοιο μέτρο που εκ των πραγμάτων μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμούς, στέρηση της ελευθερίας, είναι οδηγήσει σε περιορισμούς. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση ούτως ή άλλως πρέπει να λειτουργεί κανονικά η εφαρμογή των εγγύσεων της οδηγίας. Τώρα θα σας πω κάτι που δεν περιλαμβάνεται στις πτυχές που εξετάζονται από την οδηγία, αλλά προσέξτε, μερικές φορές το να αναφέρουμε παιδευτικές δραστηριότητες, τέτοιου είδους παρεμβάσεις που περιορίζουν σε κάποιο βαθμό την ε, προσωπική ελευθερία, ακόμα και αν αλλάζουμε τα όρια, τα ηλικιακά, αυτά τα age thresholds, τα ηλικιακά κατόφλια for liability to prosecution, δηλαδή ηλικιακά όρια για να διωχθεί κάποιο ποινικά, πρέπει να προσέχουμε ε, αυτή η ετικέτα που επικαλάμε να μην μεταβληθεί σε παράκαμψη της ουσιαστικής εγγύησης. Κατά την άποψή μου λοιπόν οι εγγύησεις της οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις υποθέσεις που μπορεί να συνεπάγονται εφαρμογή περιοριστικών μέτρων ή αρνη και σε επιπτώσεις για τον ανήλικο που μπορεί να είναι μέτρα μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη της προσωπικότητας ή μέτρα που παρότι δεν περιλαμβάνουν την επίσημη, μια επίσημη ποινική κύρωση μπορεί ούτως ή άλλως εγγενώς να περιλαμβάνουν κάποια επιβεβαίωση ευθύνης δηλαδή εναλλακτικά μέτρα που αντικαθιστούν την καταδίκη και τα οποία ακόμη και αν οδηγούν σε στέρηση της προσωπικής ελευθερίας ε, αποδίδουν κάποια ευθύνη. Επίσης τώρα τα δικαιώματα των ανηλίκων ε, και η ατομική αξιολόγηση. Η ατομική αξιολόγηση είναι θεμελιώδη σημασία ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή οποιασδήποτε απόφαση έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια της, της διαδικασίας και στο πέρας της διαδικασίας ώστε να διασφαλίζει όπως είπα μία πραγματικά προσαρμοσμένη στο άτομο απόφαση. Απόφαση δηλαδή που θα προσαρμόζεται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ανηλίκου. Γι' αυτό το λόγο το άρθρο 7 της οδηγίας το οποίο παρότι δεν διευκρινίζει συγκεκριμένα τους σκοπούς αυτής της ατομικής ε, αξιολόγησης, πρέπει να επιτρέπει την επιλογή των διαφόρων ε, ρεαλιστικών επιλογών είτε κατά τη διάρκεια είτε στο πέρας της διαδικασίας. Συνεπώς ακόμη και αν δεν έχουμε καταλήξει μια τελική απόφαση που επιβεβαιώνει την ευθύνη, ακόμη και η εφαρμογή ενός προστατευτικού μέτρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια απαραίτητα ατομική αξιολόγηση του κατηγορουμένου. Κάτι άλλο σημαντικό, τα δικαιώματα του ανηλίκου πριν από την ε, δίκη. Αυτό σχετίζεται με την ιδέα ότι για τον ανήλικο η δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του εξαρτάται από την ικανότητά του να κατανοήσει και να συμμετάσχει συνειδητά στη διαδικασία. Η παρουσία του δηλαδή μαζί με μια σειρά άλλων εγγύσεων που προβλέπονται στη διαδικασία αποτελούν ε, απαραβίαστες συνθήκες ε, όχι μόνο για τον ενήλικο. Επαναλαμβάνω, η παρουσία του ανηλίκου στη διαδικασία είναι πολύ σημαντική και για τον δικαστή. Διότι συχνά η παράσταση του ανηλίκου μπορεί να παράσχει στο δικαστή συγκεκριμένες ενδείξεις οι οποίες δεν είναι διακριτές ε, στις αξιολογήσεις προσωπικότητας. Είναι απολύτως σημαντική η αναφορά στο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις ατομικές αξιολογήσεις τους ανηλίκους οι οποίοι εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες που εξανακάζονται να εκτελέσουν κάποια πράγματα ως θύματα της διακίνησης ατόμων. Να υπενθυμίσω ότι σε πολλές περιπτώσεις εδώ έχουμε ανηλίκους δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ τις συνέπειες που έχει μετανάστευση σε τέτοια ανήλικα άτομα που τα ε, θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο να συμμετάσχουν σε κλιματικές διαδικασίες ή να υπάρξουν θύματα αυτών. Το δικαίωμα προστασίας της γονικής ευθύνης. Το να ερμηνεύεται κανείς για τα δικαιώματα του ανηλίκου, αυτό είναι το άρθρο 5 και παράσταση στην ακρόαση, αυτό είναι το άρθρο 15. Αυτές είναι δύο διατάξεις οι οποίες αναφέρονται σε δύο πράγματα. Από τη μια υπάρχει απέτηση ότι θα πρέπει ο γονιός να γνωρίζει ακριβώς όσα διαπιστώνονται και να βρίσκεται δίπλα στον ανήλικο στις διάφορες επιλογές που θα κάνει αλλά και να βοηθήσει ψυχολογικά με αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό τον λόγο, όταν μιλάμε για τον ε, ιδανικό ε, ενήλικα που μπορεί να αντικαταστήσει τον γονιό, θα πρόσθετα την ε, φράση που υποδεικνύεται βάσει επιλογής του ανηλίκου. Τώρα, όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης στον κηδεμόνα, ε, αυτός βεβαίως συμφωνώ θα πρέπει να ενημερώνεται κατά την άποψή μου δεν προβλέπεται και θα έπρεπε μια υποχρέωση ειδοποίησης της, για την ακρόαση και σε κάποιο μέτρο θα πρέπει να επιβάλλεται κύρωση σε περίπτωση τέτοιας, ε, απουσίας τέτοιας προειδοποίησης. Γενικά πολλές από τις εγγύησεις της οδηγίας δεν περιλαμβάνουν κύρωση σε περίπτωση παραβίασης. Τελευταίο πράγμα, υποχρεωτική παράσταση του εναγωμένου. Ναι, πάντα σε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Να μην προβλεφθούν περαιτέρω εξηγήσει. Όλα τα σενάρια στα οποία εφαρμόζονται στα οποία εφαρμοστεί η οδηγία πρέπει να γίνονται με παρουσία του ανηλίκου. Και τελευταία υποχρέωση συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μέτρα. Δεν ε, θα συνεχίσω άλλο, βλέπω ότι έχει λήξει ο χρόνος μου. Εκπαιδευτικά μέτρα συμπληρωματικά ή εναλλακτικά σε σχέση με τυχόν προστατευτικά μέτρα ή κυρώσεις. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εάν δεν έχει επιβεβαιωθεί η ευθύνη, δεν μπορούν ε, τα παιδευτικά συστήματα να λάβουν ε, υπό την προστασία τους, υπό την ευθύνη τους ε, κάποιο ύποπτο κατηγορούμενο άτομο. Ευχαριστούμε την κυρία Πατανέ που μας παρήχε πολύ σημαντικές πληροφορίες δικαστικού χαρακτήρα, πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστούμε την καθηγήτρια την κυρία Σαπατανέ. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ε, να δώσω το λόγο στους συναδέλφους γιατί μέσω των ερωτήσεών τους μπορούμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω το θέμα που εξετάζουμε. Δίνω λοιπόν το λόγο στην συνάδελφα την κυρία Σάκη για την ερώτησή της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τους ομιλητές για την ηλικία της ποινική ευθύνη. Η πρόταση της οδηγίας αναφέρει τα 18 έτη. Το ανώτατο αυτό όριο έχει τεθεί παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν θέσει τα 17 έτη ως ανώτατο όριο για τα δικήματα ανηλίκων. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν επιθυμεί να ασχοληθεί, να αλλάξει την ηλικία της ποινική ευθύνης παρά τις διαφορετικές πρακτικές των κρατών μελών. Σε πολλά κράτη-μέλη το όριο είναι 14 ή 15 ε, χρόνια και μόνο 5 κράτη-μέλη έχουν χαμηλότερο όριο ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω τους ειδικού μας για το αν υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης του ορίου ηλικία της ποινική ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη τι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με τη σημασία της εναρμόνισης ε, της αξιολόγησης των ανηλίκων, οι οποίοι δεν έχουν τα ε, κατάλληλα έγγραφα πάνω τους. Αξιολόγηση της ηλικία λοιπόν των ανηλίκων πολλές φορές είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ωστόσο, εάν έχει εκτιμηθεί η ηλικία του ανηλίκου παραπάνω από όσο είναι, ο ανήλικος μπορεί να μην έχει την κατάλληλη προστασία. Τι γνώμη έχουν λοιπόν οι εμπειρογνώμονές μας για την ανάγκη της εναρμόνισης του καθορισμού του ορίου ηλικία ενό ανηλίκου. Έχουμε ακόμα μια ερώτηση. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και αυτή την άλλη ερώτηση και μετά οι εμπειρογνωμονές μα μπορούν να απαντήσουν και στι δύο ερωτήσει. Το λόγο λοιπόν έχει συνάδελφο Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, εμπειρογνώμονές μας. Η ερώτηση μου σχετίζεται με την κράτηση η οποία η κράτηση ανηλίκων είναι διαφορετική από την κράτηση ενηλίκων. Από αυτά που βλέπουμε λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς ορίζουμε ή πώς καθορίζουμε το όριο ηλικία. Αν θεωρήσουμε ότι τα 18 είναι το όριο ηλικία, ε, όριο ηλικίωση μάλλον, θα πρέπει να δούμε και τον ορισμό των. Ε, των μικρών αδικημάτων. Και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά σε κάποιο νέο άνθρωπο, εάν αυτά δηλαδή έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην μελλοντική ζωή του, αν θα πρέπει να καταγράφονται. Και τέλος, εάν έχετε κάποια σχόλια ε, για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο κείμενο του Συμβουλίου και στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη συμμόρφωση του Συμβουλίου στις ε, καλές πρακτικές και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα μια ερώτηση από την κυρία Βόζενμπεργκ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω για τις εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες που πήραμε σήμερα από τους διακεκριμένους ομιλητές. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον θα έπρεπε να μας προβληματίσει και η ηλικία των δραστών όταν είναι ανήλικοι σε αξιόπινες πράξεις τις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα τα οποία και με την ιδιότητα του δράστη και με την ιδιότητα του θύματος είναι ανήλικοι. Και επίσης ε, γνωρίζετε ότι στα κράτη-μέλη υπάρχει διαφορετική μεταχείριση, ποινική μεταχείριση για συγκεκριμένες πράξεις σε ανηλίκους ανάλογα με την ανηλικότητα. Δηλαδή διαφορετικά τιμωρείται ένας ανήλικος 10 ετών για, την, για μία και συγκεκριμένη πράξη, διαφορετικά αν είναι 12, διαφορετικά αν είναι 14. Τουλάχιστον στη χώρα μου στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η διακύμανση και από ό,τι ξέρω και σε άλλα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό θα μπορούσε να οριοθετηθεί έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή μεταχείριση σε σχέση με τους ανηλίκους και σε σχέση με την παρατήρηση που έκανε η κυρία δικαστής για το συμφέρον του ανηλίκου. Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι εξαιρετικά όριστη η έννοια και εναπόκειται στην κρίση του δικαστή. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό σωστά οριοθετείται γιατί ο δικαστής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και στο να κρίνει καθοριστικά το συμφέρον του ανηλίκου. Αλλά βλέπουμε περιπτώσεις περιπτώσεις όπου παραδείγματο χάρη στον τομέα της μεταναστεύσεως όπου δεν είναι πολλές φορές ε, στους ανήλικους δεν είναι διακριτή η ανηλικότητα. Μπορεί ένας ε, να δηλώσει μια άλλη, μια ψευδή ηλικία και εκεί να μην μπορεί να διακριθεί ε, κατά πόσο είναι υπεύθυνο, σε ποιο βαθμό είναι υπεύθυνο, είναι τελικά ανήλικος ή θα πρέπει να τον μεταχειριστεί το δικαστήριο και στο ανακριτικό στάδιο, οι ανακριτικές αρχές και μετέπειτα στη δίκη αν προσδιοριστεί σε χρονικά πλαίσια που να εντάσσονται μέσα στην απόκληση αυτή ως ενήλικο. Αν αυτά μας έχουν απασχολήσει, φαντάζομαι είναι πολύ δύσκολη η οριοθέτηση, αλλά μπορούμε να συμβάλλουμε με κάποιες απόψεις που να βοηθήσουμε στον προβληματισμό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους και δίνω τώρα το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα πέντε λεπτά ο καθένας. Ακολουθούμε την ίδια σειρά παρεμβάσεων. Το λόγο έχει ο Δ. Πιγκάλ. Oui, euh, je vais Λοιπόν, θα ξεκινήσω τις απαντήσεις μου. Σε ό,τι αφορά την ηλικία ποινική ευθύνη η εντολή της Κομισιόν ήταν ακριβώς να μην υπάρχει ε, αλλά όπως υπενθυμίσατε υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο λένε ότι μέχρι τα 18 το θέμα είναι να λαμβάνονται μόνο εκπαιδευτικά μέτρα, αν και από τα 16 και μετά θα μπορούσε ο νέος να δικαστεί από ένα δικαστήριο ενηλίκων και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα και απ' την άλλη έχουμε χώρες όπως το Ενωμένο Βασίλειο, 10 χρόνια νομίζω είναι το επίπεδο, ίσως και πιο χαμηλό, από τα 7-8 χρόνια είχαμε μια πολύ γνωστή υπόθεση από κάποια χρόνια, θα τη θυμάστε. Άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά 7 έως 10 από τη μία και 18 από την άλλη. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν ήθελε να μπει σε αυτά τα χωράφια, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσει ε, κάποια συνεκτικά μέτρα, γιατί υπάρχουν διαφορετικά νομικά συστήματα, διαδικασίες, ε, εκπλοκισμός Βέβαια, επιθυμητό θα ήταν και ευκταίο να υπάρχουν κάποια κατώτατα όρια ηλικιακά. Ένα παιδί 10 ετών δεν είναι το ίδιο με έναν έφηβο 17 ή 17 μισό. Και παίρνω το παράδειγμα της Γαλλίας για τους ανηλίκους. Κατά από τα 13, ένας ανήλικος δεν μπορεί να καταδικαστεί να του επιβληθεί μια ποινή. 10-13. Σε, αυτά, σε αυτές τις επιβάλλονται μόνο εκπαιδευτικά μέτρα. Υπάρχει όμως και μια άλλη όροφη, ένα σκαλοπάτι από τα 13 στα 16 χρόνια. Εκεί ο ανήλικος έχει ένα ελαφρυντικό ε, λόγω της ηλικία του και αν καταδικαστεί από ένα δικαστήριο δεν θα του επιβληθεί η ίδια ποινή με αυτή που θα επιβάλλεται σε έναν ενήλικο. Και έπειτα έχουμε το, 16, το ηλικιακο όρο 16-18, που και πάλι μπορεί να είναι ελαφρυντικό το ανήλικον, ε, αλλά μπορεί να το επιβληθεί παρόλα αυτά, το δικαστήριο διαλέγει την ποινή. Λοιπόν, θα προσπαθήσω εκτός μικροφώνου για μιλήτρια. Λοιπόν, να δώσω απαντήσεις ε, στα όσα ρωτήσατε το πρόβλημα του ορίου ηλικίας ποινική ευθύνη. Εκ των πραγμάτων το πρόβλημα αυτό αποτελεί αγκάθι για την ομογενοποίηση των εγγύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάθε χώρα έχει κάνει τις επιλογές της. Όπως είπαμε, η πρόταση οδηγίας δεν ασχολείται με τα ηλικιακά όρια, από επιλογή. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα κατά με. Γιατί διότι δεν είναι ο ορισμός επίσημα του ορίου μέγιστης και κατώτης ηλικία. Ε, το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε ενώπιον ενός ε, ανηλίκου που είναι κάτω από την ελάχιστη ηλικία. Εάν εγώ ορίσω την ηλικία ποινική ευθύνη στα 14 έτη και μετά επιτρέψω μέσω μέτρων επίσημα μη ποινικών να περιοριστεί, να στερήσω την ελευθερία ενός ατόμου επικαλούμενος ε, πανεκπαίδευση, παρέμβαση προς κάποιο άτομο το οποίο δεν μπορεί να καταδικαστεί εκεί τίθεται το πρόβλημα των εγγύσεων για το μέγιστο όριο 18-17 ετών και εκεί υπάρχει μια τάση και το λένε πολλοί διεθνείς χάρτες να ορίζεται ανήλικος ε, κάποιος ο οποίος βρίσκεται λίγο κατά από τα 18. Μάλιστα στην οδηγία αναφέρεται ότι οι εγγυήσει ε, εφαρμόζονται στην ηλικία του ανηλίκου από τη στιγμή που έχει οριστεί ως ύποπτος κατηγορούμενος. Αυτό είναι κριτήριο για να τεθεί σε λειτουργία η οδηγία. Άλλες χώρες ορίζουν στις εθνικές τους νομοθεσίες ότι το εν λόγω άτομο εντάσσεται σε δικαιοδοσία ανηλίκων από τη στιγμή που έχει διαπράξει το έγκλημα. Δηλαδή η στιγμή που διαπράχθηκε το έγκλημα ορίζει το κατά πόσο δεν σε ισχύει αυτές οι εγγύσεις. Όσον αφορά την αποτελεσματική μεταχείριση ενός ανηλίκου του οποίου την ηλικία δεν μπορούμε να επικυρώσουμε. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Στην Ιταλία, για να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, αν και μόνο ενδεικτικό, υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του ανηλίκου συνεργατικά, δηλαδή πρέπει να παράσχει στοιχεία. Εάν αυτά δεν είναι αξιόπιστα, πέραν των δακτυλικών αποτυπωμάτων που πάνε να και τα συγκρίνουμε με τη Διεθνή Βάση Δεδομένων Άφης, εκεί υπάρχει δυνατότητα να εξεταστεί ένα δείγμα οστών και σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται δεδομένη η ελάχιστη ηλικία. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει βεβαιότητα θεωρούμε δεδομένη την ελάχιστη ηλικία. Το τελευταίο τώρα όσον αφορά το ποια μπορεί να είναι μεταχείριση των νέων ενηλίκων. Ε, η κατηγορία των νέων ενηλίκων είναι επικοινόμορφη και αυτή σε κάθε χώρα είναι διαφορετική. σε κάποιες άλλες, ε, σε κάποιες επεκτείνεται η κατηγορία των ανηλίκων, σε άλλες των ανηλίκων, ανηλίκων, σε άλλες υπάρχει ειδική κατηγορία. Το βασικό στοιχείο είναι η ειδική μεταχείριση, το καθεστώς ενισχυμένων εγγυήσεων, είτε λόγω του γεγονότος ότι τα άτομα αυτά έχουν διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκημα, ή είναι ανακρινόμενοι σε μια διαδικασία όταν ήταν ανήλικοι. Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση στην απόφαση θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτή τη συνθήκη, στην ευάλωτη συνθήκη στην οποία βρισκόταν το άτομο όταν διαπράξει το έγκλημα. Θα διακόψω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πατενέ και τον Δ. Πικάλ για τις περαιτέρω διευκρινήσεις μας εδώ σαν ερωτήσεων να σε ευχαριστήσω και πάλι όλους και ξαναδίνω τώρα το λόγο στον Πρόεδρο τον κύριο Μωράς για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Κατρίνα. Παίρναμε τώρα στο δεύτερο πάνελ για τη νομική συνδρομή, στο οποίο θα προεδρεύσει ο Ντένις Τε ο οποίος είναι και ο εισηγητής της ιετικής έκθεσης. Θα ήθελα επίσης να καλέσω και τους επιρρογνώμονες, τον Εμίλιο Αλβάρες Αλτσέδο και τον κύριο Ζάζαν Ναμοράτζε να έρθουν στο Προεδρείο. για να αρχίσουμε. Uh, Dennis de Jong is going to take the chair for this session. Dennis. Ο Ντένις Διόγκ θα προεδρεύσει σε αυτό εδώ το τμήμα της συνεδρίασης. Ντένις, έχεις το λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλοντ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι είστε ακόμα ξύπνοι και δραστηροί. Θα προσπαθήσω λοιπόν να επιταχύνω λίγο τη διαδικασία, διότι νομίζω πως έχουμε αργήσει 8 με 10 λεπτά. Έχουμε έρθει εδώ για να ακούσουμε σημαντικούς ανθρώπους, τους οποίους καλέσαμε για να μας βοηθήσουν στο έργο μας. Γι' αυτό λοιπόν θα περιοριστώ αφού μιλήσουν οι εμπειρογνώμονε μα και δεν θα μακρηγορήσω για την έκθεσή μου. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Εμίλιο Αλβαρέ Σαλσέδο, από το Υπουργείο Δικαιοσύνη τη Ισπανία, ο οποίο θα είναι ο πρώτο ε, ομιλητής τώρα. Έχετε το λόγο. Muchas por... Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για την πρόσκληση που απευθύνεται στην Ισπανία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο και εκπροσωπώ. Θα σας μιλήσω για το ευεργέτημα παινία στη δωρεάν δικαστική αρρωγή και θα σας περιγράψω το σύστημα που έχουμε στη χώρα μου, στην Ισπανία. Καταρχάς όμως να σας πω ότι κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ισπανίας ε, ε, το σύστημα το ισπανικό για τη δωρεάν ε, παρογή, νομική αρρωγής είναι από τα πιο γενναιόδωρα ε, και ευρύτατα που υπάρχουν, διότι καλύπτει όλα τα επίπεδα της ένωμης τάξης και όχι μόνο τους υπηκόους της Ισπανία ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιασδήποτε άλλης χώρας που διαμένουν νόμιμα στην Ισπανία, καλύπτει όλους τους πολίτες που για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται σε ισπανικό έδαφος. Το ευεργέτημα παινία στην Ισπανία είναι πυλώνα του δικαστικού συστήματος, γιατί ε, παρέχει δωρεάν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στους πλέον ευαίσθητους και στα πιο ε, μειονεκτούτα ε, στρώματα. Έχουμε το άρθρο 24 και 25 του συντάγματος που ε, είναι το επιστέγασμα της παροχής βοήθειας από το κράτος δικαίου. Αυτά τα λέει το σύνταγμά μας. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι συνταγματικές αρχές, απ' την άλλη θέλουμε όμως να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και έχουμε και γι' αυτό το άρθρο 119 του συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι είναι δωρεάν η δικαιοσύνη όπως προβλέπει ο νόμος ε, και ιδίως για όσους δεν έχουν επαρκείς πόρους ε, για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Άρα έχουμε όπως καταλαβαίνετε, ένα σταγματικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει ε, το να παρέχει ε, τις υπηρεσίες αυτές στο κράτος, ώστε να μπορεί το δικαίωμα αυτό στη δωρεάν δικαστική ε, αρρωγή να είναι εξασφαλισμένο για οποιονδήποτε. Και βέβαια εκπληρώνουμε όλα τις υποχρεώσεις μας και όλες τις διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω, ήθελα να σας πω... Okay. Okay en el Υπάρχουν κάποιες ομάδες, ε, έχουμε τους τροφίμους σοφρανιστικών ιδρυμάτων, ε, γυναίκες που είναι θύματα οικογενικής βίας, ε, ξένοι μετανάστες, που αυτοί πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη και οι δικηγόροι, οι νομικοί παραστάτες. Το μοντέλο μας είναι πολύπλοκο, γιατί το Ισπανικό κράτος είναι πολύπλοκο Έχουμε τη γενική διοίκηση και έχουμε και τις αυτονομίες, τις αυτόνομες περιφέρειες. Ε, και το Ευρύτερο παινίας παρέχεται στην Ισπανία από το κράτος σε πέντε αυτόνομες περιφέρειες ε, που ακόμα ε, δεν έχουν μεταφέρει αυτά τα και στις 12 δια ε, αυτόνομες περιφέρειες οι ίδιες αυτές διαχειρίζονται αυτό το ευεργέτημα παινίας. Μπορεί ο νόμος να είναι, απέναντι στον νόμο να νολίσει, δεν είναι όμως ίδια, ε, ίδιες οι νομικές ρυθμίσεις σε όλες τις ε, αυτόνομες ε, περιφέρειες. Έχουν διαφορετικές διατάξεις αυτόνομες περιφέρειες σε πολλές περιπτώσεις. Μπορεί δηλαδή να την ίδια υπηρεσία από κάποιο δικηγόρο, αλλά να πάρει άλλη αμοιβή, ανάλογα με το σε ποια αυτόνομη περιφέρεια βρίσκεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα ο δικηγόρος υπεράσπισης. Η κατάσταση αυτή λοιπόν είναι στην Ισπανία. Δεν είναι φτηνή η ε, δικηγόρη. έχω κάποια στοιχεία για το τελευταίο έτος, το κόστος ε, επίσης του ευεργετήματος παινίας ανέρχεται σε 223 εκατομμύρια περίπου. Και παρεσχέθησε 1.774.000 άτομα. Για την οδηγία τη συγκεκριμένη, επειδή μιλάμε για ποινικό δίκαιο εδώ, η νομική παράσταση σε κρατουμένους κόστησε 44.700.000 και παρασχέθηκε σε 667.000 άτομα. Το δικαίωμα ποινία. Θα, ε, θέλω τώρα να αναφερθώ στη δομή του Ισπανικού συστήματος Τέσσερις είναι βασικοί πυλώνες. Υπάρχει, υπάρχουν 39.000 εθελοντές και εκ παρέχουν ε, τις ε, υπηρεσίες τους. Και βέβαια η υπηρεσία παρέχεται σε όποιον τη ζητήσει. Ένας άλλος πυλώνας. Είναι η οικογενειακή βία. Ε, βία ε, κυρίως κατά γυναικών. παντού στην Ισπανία υπάρχει τουλάχιστον ένας ειδικό ε, συνήγορος για αυτές τις γυναίκες. Και το τρίτο είναι ο πυλώνας αυτής της ε, οδηγίας. 365 ημέρες το χρόνο 24 ώρες την ημέρα υπάρχει τουλάχιστον ε, ένας δικηγόρος ο οποίος ε, κατά κάποιο τρόπο είναι συνεχώς στη διάθεση των ε, όσων σε αυτούς που θα χρειαστεί. Και υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι δικηγόροι που θα πρέπει βέβαια και να χρηματοδοτηθούν με κάποιο τρόπο. Το ευεργέτημα πενέσει στην Ισπανία. Δεν καταβάλλεται από το κράτος Υπάρχουν επαγγελματικέ ενώσει, οι δικηγορικοί σύλλογοι ουσιαστικά που το παρέχουν. Αυτού πληρώνει κανεί. Και αυτό γίνεται με τη μέθοδο τη επιδότηση, τη επιχορήγηση των δικηγορικών συλλόγων. Γίνεται ανατρίμηνο και σε αυτόνομε περιφέρειες και σε επίπεδο γενικής κρατικής διοίκηση, ανάλογα με τα έξοδά του. και πρέπει βέβαια να δικαιολογηθούν, ε, να αιτιολογηθούν αυτά τα έξοδα, αυτές οι δαπάνες. Με παροχή συμβουλών εσωτερική και εξωτερική. Διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας την οδηγία, προέκυψε κάτι που εμένα δεν μου είναι πολύ ξεκάθαρο. Ε, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι επειδή σε όλες τις χώρες της Ένωσης έχουμε τόσο διαφορετικά συστήματα για την παροχή του ευεργετήματος παινίας, το να προσπαθήσουμε να ομοιογενοποιήσουμε την οδηγία αυτή κάποια θέματα, μπορεί να είναι δύσκολο εγχείρημα. Ένα θέμα είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που έχει οικονομικό κόστος, αλλά και όχι μόνο οικονομικό, και διοικητικό κόστος και κόστος διαχείρισης οι βουλευτές, οι εμπειρογνώμονες πρέπει να σκεφτούν αυτό το κόστος. Όλοι όσοι εξεργάζονται αυτή την οδηγία. Δηλαδή τελικά ποια είναι τα πλεονεκτήματα τελικά αυτού του ευρωπαϊκού εντάλματος. Δεν ξέρω ποιος εκδίδει τέτοια εντάλματα και ποιος είναι αποδέκτης, αλλά κάπως πρέπει και να χρηματοδοτηθούν. Αν η Ισπανία δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το κρατικό κορβανά στην Ισπανία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να την πληρώσει τελικά ε, οι φορολογούμενοι. Αν ατραβήστε το μεχαρίσμα που que se considere más conveniente un sistema para θα πρέπει να ε, υπάρξει ένα σύστημα για την ε, αντιστάθμιση αυτού του κόστους. Ε, μιλάω για την Ισπανία, αλλά μπορώ να μιλήσω για οποιαδήποτε άλλη χώρα, η Πορτογαλία, δεν ξέρω. Αν εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης για τη Γαλλία, ποιος πρέπει να το, η κράτηση, ποιος πρέπει να πληρώσει η Γαλλία ή η Πορτογαλία. Αυτά όλα πρέπει να οριστούν. Υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι η στέρηση ελευθερίας. Αναφέρεται η οδηγία στο θέμα και είναι πολύ μεγάλη ε, η ανησυχία μας ε, για αυτό το ζήτημα στην Ισπανία. Αυτά τα άτομα ε, που τους έχει επιβληθεί ποινή στέρης ελευθερίας, πώς τους εξασφαλίζουμε σε αυτούς τους ανθρώπους το ευεργέτημα παινίας. Αφού δεν μπορούν να πάνε σε δικηγόρο, πρέπει ο δικηγόρος να πάει σε αυτούς. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες ε, σοφρονιστικού ε, δικηγορικού προσανατολισμού, γιατί θέλουμε και στα σοφρονιστικά ιδρύματα να πάει το ευρύτημα παινής, αλλά αυτό έχει κόστος. Πρέπει σε κάθε σοφρονιστικό ίδρυμα να συναυθούν συμφωνίες με τα δικηγορικά σωματεία, με τους δικηγορικούς συλλόγους, για να μπορούν δικηγόροι να συντρέχουν άτομα τα οποία χρειάζονται δωρεάν διακαστική αρρωγή. Και έπειτα έχουν και το θέμα των αλλοδαπών. Το ζήτημα των αλλοδαπών στην Ισπανία, που είναι μια χώρα ε, συνοριακή, με την έννοια ότι έχει τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης εκεί, έχουμε και πρόβλημα με ανηλίκους ε, που έρχονται στα σύνορα τα εξωτερικά της Ένωσης και πρέπει να τους ε, προσφέρουμε υπηρεσίες. Έχουμε τα ζητήματα της μετανάστευσης του ασύλου. Τα άτομα που φτάνουν ε, στην ε, Ισπανική επικράτεια, στα σύνορα, αμέσως δικαιούνται αυτόματα ε, την δωρεάν δικαστρική αρρωγή. Μπορεί ακόμη και κάποιος που έχει συλληφθεί από τις αρχές να δικαιούται αυτή την βοήθεια, το ευεργέτημα απενίαση είτε ανήλικο είτε ενήλικο Και αν είναι ανήλικο και ε, τις κοινωνικές υπηρεσίες δικαιούται. Αυτά ήθελα να αναφέρω, δεν ήθελα να εμβαθύνω στα διάφορα σημεία. Εν κατακλείδη όμως ήθελα να πω το εξής, πολύ σημαντικό. Η δωρεάν δικαιοσύνη έχει κόστος, κοστίζει και μάλιστα πολύ. Στην Ισπανία καταβάλλεται κάθε δυνατή δημοσιονομική προσπάθεια για να μπορεί το ευεργέτημα παινίας να παρέχεται σε όλους τους πολίτες ή μάλλον η δικαιοσύνη να παρέχεται, να απονέμεται σε όλους τους πολίτες. Είχαμε Έχουμε διαφορετικούς συντελεστές για τις αμοιβέ των δικηγόρων, έχουμε μειώσεις και πολλές φορές να πω ότι είναι ήρωες οι δικηγόροι γιατί παρότι δεν αμείβονται επαρκώς παρέχουν υπηρεσίες σε χιλιάδες άτομα που αλλιώς δεν θα είχαν πρόσβαση στην ε, δικαστική ή νομική παράσταση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω πως ήταν πολύ τιμή συνεισφορά στην σίγουρα ενδιαφέρουσα συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι μετά τον δεύτερο μιλητή θα καταστήσει ευχαριστώ αυτό. Δεύτερος ομιλητής, ο Ζάζα Εναμοράτζε, ο οποίος είναι διευθυντής μια ΜΚΟ στη Βουδαπέστη που έχει να κάνει με δικαστική συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μην μιλήσετε πάνω από 10 λεπτά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω εδώ και να σας δώσω Πληροφορίε, ε, ιδιαίτερα μάλιστα όταν συζητάτε τρει πάρα πολύ βασικέ οδηγίε που σχετίζονται με του υπόπτου στι ποινικέ διαδικασίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει πολύ τα τελευταία χρόνια να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των υπόπτων σε όλη την επικράτεια τη ε, Ένωση και αυτέ οι οδηγίε είναι το αποτέλεσμα των εργασιών τη. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω και την άποψη των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Ο δικός μου οργανισμός η Open Justice Initiative εδώ και 15 χρόνια εργάζεται στον τομέα της νομικής συνδρομής. Δραστηριοποιούμαστε στα αστυνομικά τμήματα, διασφαλίζουμε έγκαιρη και γρήγορη πρόσβαση σε νομική συνδρομή, παρέχουμε πληροφόρηση για αυτή ε, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα διασυνοριακό δίκτυο ε, συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με 18 κράτη-μέλη σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα. Στα πλαίσια αυτά, φέτος το Μάιο, μαζί με το Justice Network, διοργανώσαμε ένα συνέδριο με 40 εμπειρογνώμονες ανάμεσά τους δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου, μέλη της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη-μέλη για να αναθεωρήσουμε και να αναλύσουμε τις διατάξεις της οδηγίας που σχετίζονται με την νομική αρρωγή. Τρεις παρατηρήσεις έγιναν. Καταρχάς, αναγνωρίστηκε η σημασία της οδηγίας, ή των οδηγιών μάλιστα, και η σημαντική συνεισφορά της στη βελτίωση της κατάστασης. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν αναγκαίος και ουσιαστικός στην βελτίωση της οδηγίας. Έπειτα, η οδηγία για την νομική συνδρομή σχετίζεται άμεσα με την οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Διότι Από το 2003 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εργάζεται πάνω στα δικονομικά δικαιώματα, θεώρησε αυτό το δικαίωμα όσο βασικό και θεμελιώδες. Και αργότερα υπήρξε επιθυμία όλα αυτά τα δικονομικά ζητήματα να ρυθμίζονται από το μέτρο C, έτσι λεγόταν, από ένα ενιαίο μέτρο. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων λοιπόν διαβουλεύτηκε για τις οδηγίες και για αυτό το μέτρο C, το οποίο ήταν αρκετά αμφιλεγόμενο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποιο στάδιο ήταν να χωριστεί η οδηγία σε δύο διαφορετικές οδηγίες και έτσι προέκυψε η C1 η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα και η C2 η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή. Έπειτα, οι οργανισμοί αυτοί εξέφασαν τις ανησυχίες τους για αυτή την κατακαιρματισμένη προσέγγιση της ε, παροχής νομικής συνδρομής, διότι υπάρχει ο φόβος ότι αυτή η κατακαιρματισμένη προσέγγιση θα δημιουργήσει κενά. Χρειάζονται προτάσεις ε, και για διασφαλίσεις, διότι η πρόσβαση στην ε, σωστή και αποτελεσματική νομική συνδρομή προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη. Και αυτό ε, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο αντιμετωπίζονται προβλήματα στην Ευρώπη. Πρακτικά δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο σύστημα νομικής συνδρομής που να εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Ένα ενιαίο σύστημα. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία και το πεδίο εφαρμογής, καταρχάς. Εμείς προτείνουμε ένα πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ε, για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Έχουμε διατυπώσει την πρόταση η οδηγία αυτή να ε, αφορά μόνο όσους ε, έχουν στερηθεί την ελευθερία τους. Έπειτα, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της κατηγορίας που τους βαρύνει. Τώρα το χρονοδιάγραμμα είναι επίσης ασαφές και σύμφωνα με την οδηγία ενδέχεται κάποιος να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε νομική συνδρομή και αυτό είναι ζήτημα ορών. Πιστεύουμε λοιπόν εδώ πως το πεδίο εφαρμογή πρέπει να διευρυνθεί για να καλύπτει μια περιοχή, μια, ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι ότου ο κατηγορούμενος να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να του απαγγελθούν κατηγορίες. Η παροχή επίση νομικής συνδρομής θα πρέπει να υπάρχει μέχρι ότου ο κατηγορούμενος να χρησιμοποιήσει δικηγόρο. Η διακοπή των ε, νομικών υπηρεσιών έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην εξέλιξη της μιας υπόθεσης. Και εδώ συνδέεται και το ότι η οδηγία πρέπει να συνδέεται με την αντίστοιχη οδηγία πρόσβαση σε δικηγόρο. Υπάρχει, υπάρχουν διατάξεις για την ε, πρόσβαση σε δικηγόρο εκείνων που δεν έχουν κριθεί επιλέξιμοι για αυτό. Πρέπει λοιπόν να γίνει αναθεώρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας σε όλα τα στάδια της ε, ποινική διαδικασίας. διότι μπορεί να επηρεαστεί η επιλεξιμότητα ενός υπόπτου για νομική συνδρομή. Υπήρξε λοιπόν μία σύσταση η αποζημίωση του κόστους να μην συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και όλοι οι εμπειρογνώμονες. Έχουμε παραδείγματα προβλημάτων όπου η αστυνομία τακτικά ορίζει δικηγόρους οι οποίοι δεν είναι απόλυτα κατάλληλη. Επίσης, τη ζητήματα παροχής ε, των υπηρεσιών. Βάσει μελετών έχει προσδιοριστεί σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας και η νομική συνδρομή ουσιαστικά παρέχεται από μαθητευόμενους δικηγόρους. οι μηχανισμοί μεν είναι διαφορετικοί, οπότε θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αρχή σε αυτή την οδηγία. Το τέταρτο ζήτημα που επισημάνθηκε ήταν ότι η καθοδήγηση της οδηγίας είναι καλή για το ότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κράτη-μέλη για να κάνουν τις ε, σχετικές ε, δοκιμές και ελέγχους. Σε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σύστημα αυτό ε, που υπάρχουν περιορίζουν την πρόσβαση στη νομική συνδρομή σε πολλές χώρες. Το οικονομικό κατόφλιο για την πρόσβαση στη συνδρομή είναι τόσο χαμηλό που πολλοί αρνούνται τη νομική συνδρομή. Σε πολλές χώρες αυτό ανέρχεται στο 95%. Υπάρχουν χώρες όπου μόνο το 10% των εναγωμένων ε, έχουν δικαίωμα για νομική συνδρομή. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι κλειδί είναι η διαχείριση των νομικών υπηρεσιών. Σε ελάχιστε χώρε υπάρχει νομοθεσία νομική συνδρομή ή απαραίτητη νομοθεσία ή απαραίτητοι οργανισμοί πολύ συχνά. Υπάρχει κατακαιρματισμένη παροχή υπηρεσιών ad hoc με ελάχιστη διαχείριση επίβλεψη. Σε κάποιε χώρε ακόμη τα πιο ευαίσθητα δεδομένα δεν συλλέγονται Συνεπώ συχνά ελάχιστα γίνεται κατανόητο το πραγματικό πρόβλημα με τη νομική συνδρομή και τι επιπτώσει τη. Ούτε η οδηγία ούτε οι σύσταση περιλαμβάνουν απαιτήσει που είναι για αυτή την πρακτική και σημαντική πτυχή τη νομική σύνδρομή. Ένα από τα σημαντικά ερωτήματα για όσου χαράσουν πολιτική σε εθνικό επίπεδο είναι κατά πόσο παρέχονται κατά οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο οι υπηρεσίε αυτέ. Στο περίοδο 2000-2004 μελετήσαμε ένα νέο νομικό σύστημα το οποίο βασίστηκε σε αυτό. Ξόδευε πολλά χρήματα η κυβέρνηση στο σύστημα νομικής συνδρομής το οποίο λειτουργούσε ανεπαρκώς. Χωρίς διαφάνεια, διότι κανείς δεν είχε καμία ευθύνη γι' αυτό. Η λιθωνική κυβέρνηση έκανε μεταρρυθμίσεις και όρισε συγκεκριμένο δημοσιο οργανισμό για την οργάνωση της ε, νομικής συνδρομής. Το ίδιο συμβαίνει και στις κατοχώρες. Υπάρχει ανεξάρτητος ε, οργανισμός. Ενώ ο μηχανισμός ορίζεται από το κάθε κράτος μέλος, η οδηγία θα πρέπει να απαιτεί να καθιερωθεί ένα αυτόνομο σύστημα που θα παρέχει αυτονομία και νομιμότητα της νομικής συνδρομής. Αυτές είναι οι βασικές πτυχές που προκύπτουν από τη συνάντησή μας Ευχαριστώ να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες και πρακτικά παραδείγματα. Ήδη εκπονούμε μικρές ε, περιλήψεις, ε, μονοσέλιδες για την κατάσταση της νομικής συνδρομής σε επιλεγμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δείξουμε με παραδείγματα τη φύση των προβλημάτων και να δούμε ποιες καλές πρακτικές ε, προκύπτουν. Συνεργαζόμαστε στενά με το Κοινοβούλιο δεδομένων των δύσκολων διαπραγματεύσεων για την οδηγία πρόσβαση δικηγόρο και έτσι μπορέσαμε να υιοθετήσουμε μια ισχυρή οδηγία. Χωρίς μια ισχυρή οδηγία περινομικής συνδρομής τα πρακτικά προβλήματα δεν θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και η πρόταση της Κομισιόν δεν θα διορθώσει τίποτα. Το κόστος της μη εξασφάλισης νομικής συνδρομής είναι υπερβολικό όχι μόνο για τα άτομα και για το δικαίωμα του σε δίκαιη αλλά για το σύνολο του συστήματος. Ευχαριστώ. Thank you very much. And I also thank... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι τις 5 για κάποιες ερωτήσεις. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις, Θα θέλω να πω δύο λόγια και για την έκθεση που συντάσσω. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι και ο κύριος Άλβαρης το ανέφερε. Έχουμε εδώ έναν οδικό χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα και εγγύησεις, επειδή τα κράτη-μέλη ήθελαν το ευρωπαϊκό αντέλεμα σύλληψης. Το συζητήσαμε ήδη την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δεν έγινε τίποτα όμως μέχρι τότε, ούτε από την Κομισιόν, ούτε από το Συμβούλιο και δεν μα ικανοποιεί καθόλου το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη. Αν όμως θέλετε και επιμένετε, πρέπει και εσείς να προβείτε σε κάποια ε, μέτρα για το ευεργέτημα παινίας, τη νομική συνδρομή. Δεύτερο, καθαρά από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κόστος πράγματι είναι μεγάλο, όμως εδώ βλέπουμε τις απαρχές, κάτι που θα μπορούσε να είναι μια εγγύηση για όλους όσους μπορεί να καταλήξουν να δικάζονται σε κάποια άλλη χώρα ή να διώκονται σε κάποια άλλη χώρα. Και δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια περιοριστική προσέγγιση. Νομίζω ότι το παιδί εφαρμογή τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Δεν μπορούμε ε, να περιοριστούμε σε υποθέσεις, ε, σε, σε διάφορες μόνο περιπτώσεις που έχει να κάνουν, έχουν να κάνουν μόνο με τη στέρηση ελευθερίας. Αν δεν έχουμε το πλήρες ε, πεδίο εφαρμογή της δωρεάν νομικής δρομής, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Πώς θα έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη σε δικαιοσύνη, αν δεν πάμε μέχρι τέλους. Το Συμβούλιο όμως κάνει το αντίθετο περιορίζει ακόμη περισσότερο το πεδίο εφαρμογή. Και αν δεν έχουμε πρόοδο στα θέματα αυτά σε δωρεάν ε, δικαστική ε, αρρωγή, και επειδή έχουμε και το θέμα των παιδιών, συζητήσαμε την οδηγία για τα παιδιά, αλλά και γενικότερα. Πρέπει να πω ότι θα υπάρξουν μεγάλες επιπτώσεις και για τη δική μας δουλειά στον τομέα της αμοιβαία αναγνώριση. Δόθηκαν παραδείγματα και από άλλους για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους. Και αν είμαστε περιορισμένοι και έχουμε μια περιοριστική προσέγγιση για το ευρύτημα πενίας τι μπορούμε να περιμένουμε. Σε καμιά μια μισή εβδομάδα ε, να περιμένετε μια αρκετά επιθετική έκθεση, ε, να το ξέρει το Συμβούλιο. Βέβαια πάντοτε μπορούμε να έχουμε διάλογο, να έχουμε διαπραγματεύσεις, όμως νομίζω ότι επειδή έχουμε ένα κατακαιρματισμένο τομέα, το είπε και ο ειδικό από τη Βουδαπέστη, δεν πρέπει να έχουμε καταρχάς ένα συνεκτικό κώδικα ποινική δικονομίας και από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τη σύσταση και την οδηγία για το βλήμα ποινής. Εγώ νομίζω ότι από τη νομική σκοπιά ε, είναι πολύ κακό παράδειγμα νομοθεσίας. Θα ήθελα πολλά κομμάτια της σύστασης να περάσουν και στην οδηγία. Να δούμε αν θα συμφωνήσουμε πρώτα απ' όλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βέβαια μετά θα ξεκινήσουν και διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αλλά δεν μπορώ ούτε καν να συμμετέχω στην ακρόαση, τέλο πάντων να είμαι πρόεδρο αυτού του σκέλου, αν δεν μπω βιαστείτε επιτέλου με το θέμα του τη ποινία και να έχω μια πρόταση μέχρι το τέλο του έτου. Τώρα οι συνάδελφοι, η κυρία Σίπελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και πολλά χρόνια συζητούμε για την συνεργασία αστυνομία και δικαστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούμε να την ε, αναπτύξουμε. Και αυτό είναι καλό. Και μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας αρχίσαμε να κοιτάζουμε και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, δηλαδή τα δικονομικά δικαιώματα και αυτά φυσικά ανήκουν επίσης στα μέτρα και είναι, μια, και είναι μέτρα εξισορρόπησης ε, κατηγορούμενου και κατηγόρου. Και πρέπει επίσης να συζητήσουμε και για τις ε, οικονομικές επιπτώσεις που έχουν. Και έχω προβληματιστεί από το πόσο συχνά επαναλαμβάνεται ο όρος κόστος. Και πραγματικά έχω σταματήσει να μετράω πόσο συχνά λέμε ε, για κόστος και μου φαίνεται πως ε, αυτό είναι το σημαντικότερο. Το κόστος είναι το σημαντικότερο και όλα τα άλλα είναι δευτερεύουσα σημασίας. Και από ό,τι φαίνεται και στους άλλους τομείς και στην ποινική διαδικασία ε, υπάρχει και το θέμα του κόστους. Όμως, αυτό μου φαίνεται αρκετά ανησυχητικό και προβληματικό μάλιστα, ιδιαίτερα όταν κάνουμε λόγο για ανθρώπινα δικαιώματα, για προάσπιση δικαιωμάτων κτλ. Να μιλάμε για το πόσο κοστίζει. Και αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να εναρμονίσουμε την κατάσταση στα 28 διαφορετικά κρατημέλη. Αυτό όμω είναι και το έργο μα. Το έργο μα είναι να φροντίσουμε για μια πιο εναρμονισμένη διαδικασία έτσι ώστε να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία και να βελτιωθεί, να γίνει καλύτερη από ό,τι είναι τώρα και από την πλευρά ε, των αστυνομικών αρχών αλλά και από την πλευρά του κατηγορούμενου. Γι' αυτό λοιπόν και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι καταστήσατε σαφές ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο για πολλούς ε, ανθρώπους δεν έχει καμία ακριβώς σημασία διότι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να τον πληρώσουν. Χρειάζονται επίσης πάρα πολλές ε, διευκρινήσεις πρακτικές διευκρινήσεις. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ε, το μόνο που έχουμε να προτείνουμε σε εσάς είναι ξανά να πούμε ότι όποιος θέλει καλή συνεργασία αστυνομικών αρχών και δικαστικών να ε, επενδύσει οικονομικά σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ Πύρκη Τσίπελ. Κυρία Σαργεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά, κυρία Ζίπελ, ε, είπατε αυτά ακριβώς που ήθελα να πω. Από το στόμα μου τα πήρατε. Φαίνεται πως εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε όλη την ίδια γραμμή. Υπάρχει αρχή της αμοιβαία εμπιστοσύνη, το οποίο ήταν κάτι καινούριο που άκουσα όταν πρώτο ήρθα σε αυτό το κοινοβούλιο. Όμως, πραγματικά σκέφτομαι ότι ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας θα έπρεπε να υπάρχει συμφωνία απόψεων σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πρόκειται για τον καλό των συμπολιτών μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια βασική αρχή της κοινωνίας μας. Φυσικά, Άκουσα και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ισπανίας, ο οποίος μας ανέφερε ε, τους πάρα πολύ μεγάλους χρόνους προφυλάκησης. Επομένως, αν θέλετε εσείς να αρχίσετε να εφαρμόσετε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, πρέπει να λάβατε υπόψη και αυτές τις πτυχές, διότι αυτές οι πτυχές θα κοστίσουν πολύ ακριβά. διότι δεν θα μπορεί να καταστεί δυνατή μια περαιτέρω ενοποίηση της ε, αστυνομικής συνεργασίας στα ποινικά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και πραγματικά πιστεύω πως ε, μπορούμε να δούμε πόσο δημοκρατική είναι μια χώρα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους κατηγορούμενους και πιστεύω πως δεν επαρκούν αυτά που γίνονται τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Άλβαρες. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον δεν τα είπα καθόλου ξεκάθαρα. Γιατί μάλλον ε, σας έδωσα την εντύπωση ότι είμαι κατά της ε, αύξησης των ε, εξόδων και δαπανών για το ευεργέτημα παινίας ε, και ότι δεν πρέπει να υπάρχει δωρεάν δικαστική αρρωγή. Ετάπα πολύ άσχημα τελικά, εγώ έλεγα απλά. Ότι εμείς ακριβώς πρέπει να φροντίσουμε να παρέχεται σε όλους δωρεάν δικαιοσύνη. Αυτό είπα ότι κοστίζει πολλά χρήματα, απλά τίποτα, όχι ότι δεν πρέπει. Μακάρι μάλιστα στη χώρα μου που ξέρετε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μακάρι λέγω να είχαμε πολύ περισσότερους πόρους για να διαθέσουμε για τη δωρεάν δικαστική αρρωγή. Τα είπα χάλια, δεν τα είπα καλά. Ήθελα να σας πω ότι όχι απλά στη χώρα μας παρέχουν υπηρεσίες ε, στους υπηκόους της χώρας μου και σε άλλους υπηκόους Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αλλά όλους είπα ε, τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ισπανική επικράτεια. Όλους τους παρέχουμε αυτή την υπηρεσία του ευεργετήματος παινίας, εάν την χρειάζονται. Και είπα επίσης ότι ε, τα δεύτερα των συμπολιτών μου έχουν δικαίωμα σε αυτή την βοήθεια. Ξέρετε, έχουμε 6 εκατομμύρια ανέργου στην Ισπανία. Έχουμε 8 εκατομμύρια συνταξιούχου που παίρνουν πάρα πολύ χαμηλέ συντάξει. Οι οικογένειε τριμελής, τετραμελής, πολύ συχνά, αν ε, και οι δύο γονεί ε, είναι άνεργοι ή εργάζεται μόνο ένας, και αυτές οι οικογένειε ε, έχουν το δικαίωμα αυτό τη δωρεάν νομική αρρωγή στη χώρα μου οποιοδήποτε, είτε είναι Ισπανός, είτε υπήκος Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα. Ε, παρά τα προβλήματα που έχουμε με συγκεκριμένα σύνορα, στη Μελίγια συγκεκριμένα, σε όλα τα σύνορα που φτάνουν, που πατάνε την Ισπανική επικράτεια, έχουν δικαίωμα σε δικηγόρο για να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Αυτό είναι κάτι νομίζω, που μα βρίσκει όλου σύμφωνο. Είναι καλό. Εγώ έλεγα ότι για να παρέχουμε εξαιρετική αυτή, την εξαιρετική δωρεάν ε, ε, δικαστική αρρωγή, είπατε αυτό κοστίζει. Και δεν τα είπα καλά γιατί εγώ ίσα ίσα που είμαι υπέρμαχος ε, της ε, δωρεάν δικαστικής αρρωγής και θα ήθελα να δοθούν πόροι και μακάρι και οι δικηγόροι ε, να αμείβονταν αξιοπρεπώς όχι όπως τώρα. Και θα σας δώσω ένα στοιχείο. Οι δικηγόροι δεν έχουν ανα... Μάλλον δεν έχει αναθεωρηθεί αμοιβή τους από το 2003 και είναι ιστορική διεκδίκηση των Ισπανών δικηγόρων. Και συμφωνώ και συμμερίζομαι το πρόβλημα. Έτσι είναι όμως η χώρα μου, ξέρετε. Και ακριβώς επειδή είναι έτσι η χώρα μου όπως είναι, κάνει πάσα δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει στους περισσότερους, για να μην πω όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται, να τους παράσχει δωρεάν δικαστική συνδρομή. Σας έφερα και μια έκθεση. Ορίστε, κοιτάξτε. Από το παρατηρητήριο δωρεάν απονομής δικαιοσύνης το Υπουργείο Δικαιοσύνης που εκπροσωπώ και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συνέγραψε το έγγραφο λέει ότι η ικανοποίηση των χρηστών του ευεργετήματος παινίας είναι εξαιρετική και σας το προσφέρω. Είναι γύρω στο 90% ο βαθμός ικανοποίηση του 1,7 εκατομμύριων ανθρώπων που έχουν κάνει χρήση του ευεργετήματος παινίας στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις ε, Μεγάλη αλλαγή έχουμε στο τι είπατε και τι καταλάβαμε, ίσως ε, ωφελτε τι διαφορετικέ γλώσσες. Αλλά τώρα τα πράγματα είναι πιο σαφή. Ε, θέλατε να πείτε κάτι τελευταίο κύριε, ε, κύριε Ναμαράτζε. Χάρηκα ιδιαίτερα από τα όσα είπε ο κύριος Δεγιόγκ και τις θέσεις σας members of the Χάρηκα που άκουσα τα σχόλια των. Μου δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα η δέσμευση που έχετε για να εκπληρώσουμε αυτό το όραμα, γιατί πραγματικά όραμα είναι. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που αυτή η Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει θέση, να υψώσει τη φωνή της και να προασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών να βελτιώσουμε τις προηγούμενες οδηγίες έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Να έχουν πρόσβαση σε πραγματικά αποτελεσματική νομική αρρωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι Την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, η έκθεσή μου θα είναι έτοιμη και θα μπορέσετε όλοι να την κοιτάξετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ συνάδελφοι που ήρθατε εδώ και κάνατε δυνατή αυτή την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ σε αυτούς τους δύο καλεσμένους μας. Και πραγματικά, Ντένις, ήταν πολύ χρήσιμο το κομμάτι σου. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όσους έχουν μείνει να μην φύγουν, διότι αυτά τα τρία θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να διατηρήσουμε άσβεστο το ενδιαφέρον μας. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που έχετε δείξει ενδιαφέρον όσοι έχετε μείνει εδώ. Τέλος, η τελευταία εισηγήτρια είναι η Νάταλι Γκρίσπεκ, η οποία θα έρθει εδώ μαζί με τους Μπόστιαν Ζουπάντσικ, δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον κύριο Χόλγκερ Μάτ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου Ποινικολόγων. Και μέχρι να έρθουν θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα. Να ε, σας αρχίσουμε από τα πρακτικά ζητήματα. Έχω καταλάβει, συνάδελφοι, ότι κρυώνεται. Έτσι βλέπω. Εγώ κρυώνω τουλάχιστον. Νομίζω ότι η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Και θα επιληφθώ του ζητήματος λοιπόν, γιατί κρυώνω τόσο πολύ που επηρεάζει τη δουλειά μου. Ωραία, χαίρομαι λοιπόν που δεν είναι ιδέα μου. Θα ζητήσω να ανέβει η θερμοκρασία, γιατί Βρετανός είμαι και μ' αρέσει λίγο η ψύχρα. Και εσύ κρυώνεις Τίμωθη, έτσι. Okay. Uh, is the consensus that it's too cold? I'm just looking at all our staff members Συμφωνούμε λοιπόν όλοι πως κάνει κρύο. Να το σημειώσουμε, να το διαβιβάσουμε. Βοηθήστε με. Ωραία, θα το φροντίσω λοιπόν. Επίσης δεν με εκπλήσει ότι αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν με εκπλήσει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν καλώς έχουμε κάνει αυτή την ακρόαση. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο πάνελ και θα δώσω εδώ τη θέση μου στην Αναταλή Γκρίσπεκ για να συζητήσουμε το τεκμήριο της αθωότητας. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε όλοι. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους έμειναν, γιατί εδώ έχουμε την τρίτη σειρά παρουσιάσεων αν και αργότερα θα κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, μια πιο γενική παρουσίαση. Θα είμαι πολύ γρήγορη ώστε να μπορέσω να μπω στην ουσία του θέματος. Εισαγωγικά αυτή η δικαστική συνεργασία στο ποινικό τομέα μας βρίσκει όλους πολύ σύμφωνους και αποτελεί το αντικείμενο πολλών συζητήσεων μας επιβάλλει έναν οδικό χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων στην Ευρώπη και μας σωθεί, το λέω σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν στον προηγούμενο γερο και πιστεύω πολύ συμφωνούμε σε αυτό, μας σωθεί λοιπόν σε κάτι που επιθυμούμε όλοι να δώσουμε μια τελική μορφή σε ένα δικαστικό πλωστάσιο ευρωπαϊκού επίπεδου και όχι να έχουμε μπροστά μας ένα μοσαϊκό που αποτελείται από διάφορα διαφορετικά νομικά συστήματα των κρατών μελών, ώστε να υπάρχει κάποια μορφή αντιμετώπισης ε, των κατηγορουμένων υπόπτων στο πλαίσιο των δικονομικών διαδικασιών. Μας αποσχολούν λοιπόν εδώ τρία νομικά κείμενα τα οποία μας βοηθούν να διασφαλίσουμε ισότιμες ε, ε, διαδικασίες υπεράσπιση με τους κοινούς μας ε, κανόνες, ε, με υψηλά πρότυπα, με υψηλότερα από τα βασικά. Έχουμε μιλήσει ήδη για το τεκμήριο για το δικαίωμα παράστασης ε, στη δίκη που μας αφορά. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο ώστε να προλάβουμε να κάνουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Εδώ δίπλα μας έχουμε δύο διακεκριμένους ε, εμπειρογνώμενους, τον κύριο Ζούπαντσιτς. Ελπίζω να το έχω προφέρει σωστά. Ο οποίος ε, στη δεκάλεπτη παρουσίασή του θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του και την ανάλυση του ως δίκαστη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, σας δίνω αμέσω το λόγο για 10 λεπτά. Ε, ευχαριστώ. Merci Madame la Présidente. Je vais parler en anglais quand même. Mm-hmm. Ah, presumption of... Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Το τεκμήριο αθότητας είναι ο βασικός πυλώνας της ποινική δικονομίας. περιλαμβάνει το βάρος ε, της αποδείξεως ε, και τον κίνδυνο της μη πειθούς, ε, την αρχή του ντούπιο προωραίου που απλά σημαίνει ότι σε περίπτωση αμφιβολίας το δικαστήριο λαμβάνει απόφαση υπέρ του κατουγαρουμένου. Είναι μια παλιά ιστορία από το ρωμαϊκό δίκαιο και στο ρωμαϊκό δίκαιο έχουμε τριών ειδών τεκμήρια το πρώτο είναι το Presumptio Juris ε, που είναι απορριπταίο τεκμήριο. Το δεύτερο δεν ισχύει στο ποινικό δίκαιο από όσο ξέρω. Presumptio Juris και De Jure που είναι μη απορριπταίο τεκμήριο και μετά ε, ε η έννοια του fiction που δεν υπάρχει πια στο ε, δίκαιο, το presumption de jure de jure υπάρχει στο γαλλικό δίκαιο, όπου ένα παιδί που έχει γεννηθεί ε, ε, εντός ένα μήνου ε, αναγνωρίζει το πατέρα. Είναι κάτι πολύ εξαιρετικό στο ρωμαϊκό δίκαιο. Οι δικαστές χρειάζονταν να χρησιμοποιούν τεκμήρια σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για την υπόθεση. Διότι ο δικαστή πρέπει πάντοτε κάτι να αποφασίζει και σε περίπτωση που δεν έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται, παρόλα αυτά πρέπει να λάβει μια απόφαση. Και έτσι χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ένα τεκμήριο. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι το δίκαιο γενικότερα και επίσης και το ποινικό δίκαιο ασχολούνται με ιστορικά, όπως ονομάζονται γεγονότα, τα οποία δεν επαναλαμβάνονται εμπειρικά. Έτσι λοιπόν απόδειξη 100% στο νόμο δεν είναι δυνατή. Πάντα υπάρχει περιθώριο για εύλογες ή μη εύλογες αμφιβολίες. Στην επιστήμη μπορούμε να κάνουμε πειράματα για να αποδείξουμε κάποια γεγονότα. Αυτό δεν συμβαίνει στο δίκαιο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικά ή σε οποιασδήποτε υποθέσει από το ρωμαϊκό δίκαιο, χρησιμοποιείται το τεκμήριο. Όπως είπα προηγουμένως, στόχος ε, του τεκμηρίου, η λειτουργία του τεκμηρίου είναι να κατανείμει το βάρος της αποδείξεως και στα δύο μέρη. Και φυσικά ο κίνδυνος της ε, μη πειθούς, όπως ονομαστεί στο common law, είναι το ζήτημα του τι θα κάνει ο δικαστής σε περίπτωση εμβολίας. Με άλλα λόγια, εάν δεν τεκμηριωθούν τα αποδεκτικά στοιχεία τότε δεν κερδίζει το συγκεκριμένο μέρος της δίκης. Όπως είπα υπάρχουν δύο είδη τεκμηρίων, το απορριπταίο και το μη απορριπταίο. Ειδικότερα στην ποινική δικονομία έχουμε απορριπταίο τεκμήριο μόνο, το τεκμήριο αθότητας του εναγωμένου. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της δεύτερης παραγράφου της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το έχετε το εδώ στην οθόνη σας, οποιοδήποτε κατηγορείται με ένα ποινικό έγκλημα θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Αυτή είναι απόλυτη αρχή. Υπάρχει μία εξαίρεση, την οποία θα αναφέρω σε λίγο. Που δεν μπορεί να γίνει κανόνας. ή τα εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τώρα, δύναμη τη Ευρωπαϊκή Σύνθηξη Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, το τεκμήριο θεότητα ενεργοποιείται μόνο εφόσον έχει κατηγορηθεί ήδη με ένα ποινικό δίκημα του συγκεκριμένου άτομου. Εκεί διαθέτει το ζήτημα του ορισμού, του τι σημαίνει κατηγορία σε αυτό το τομέα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ θα μπορούσε κανεί να πει ότι ένα άτομο θεωρείται αθώο και θα πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο μεταχείρισης ως αθώος και από την αστυνομία σε προγενέστερο στάδιο. Στο Γενικό Σχόλιο 32 του άρθρου 14 τη παρέμβαση που αφορά τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα το δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2014 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΠΑ είπε όσον αφορά το τεκμήριο αθώτε είπε ότι οποιοδήποτε κατηγορείται με ποινικό αδίκημα έχει το δικαίωμα να θεωρείται αθώο μέχρι αποδείξεω του αντιθέτου σύμφωνα με τον νόμο. Το τεκμήριο αθωότητα αποτελεί θεμελιώδη στοιχείο προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβάλλει στην δίωξη το βάρο αποδείξεω. Ε, η απόδειξη πρέπει να αποδειχθεί πέραν εύλογης εμβολίας. Αυτό είναι το σκεπτικό στο οποίο βασιζόμαστε το όλο αθωότητας, η φιλοσοφία στην οποία βασίζεται, οφείλεται σε κάτι που ονομάζεται Blackstone's Ratio, αναλογία Blackstone. Επειδή προέρχεται από τα σχόλια του William Blackstone ε, επί το όνομα της Αγγλίας. Εκεί αναφέρει ότι είναι καλύτερο να διαφύγουν 10 εγκληματίες παρά να υποφέρει ένας αθώος. Αυτή είναι η βασική πολιτική στο ποινικό δίκαιο. Το τεκμήριο αθώοτας λοιπόν του εναγωμένου ή του υπόπτου. Η σύγχρονη έκδοση της ίδιας αρχής ε, είναι του Ντένις ε, στο Law of Evidence του 2007 και αναφέρει ότι το αποτέλεσμα μιας λάθος κατηγορίας θεωρείται χειρότερο κακό από την απαλλαγή. Αυτή είναι μια πολιτική που ακολουθείται στο δικαστικό σύστημα, προέρχεται από την αναγέννηση, για να το πω έτσι, και για το γνωρίζουν, εκείνη την εποχή ζούσε ο Τσέζαρ Μπεκαρία όπου στις συνθήκες του Crimes and Punishment, εγκλήματα και τιμωρίες, ε, ε, έκανε μια ρηξικέλευτη αλλαγή στα δικαστικά συστήματα της Ευρώπης, τα οποία ήταν πολύ πιο αυστηρά στη... νωρίτερα. Το ποινικό δίκαιο σήμερα περιλαμβάνει δίκες που φέρνουν σε ε, αντίθεση το κράτος και τον πολίτη και το κράτος είναι εκείνο που πρέπει να ε, φέρει, που φέρει το βάρος απόδειξης. Και αν δεν ε, υπερβεί αυτή την το απορρίψιμο τεκμήριο, τότε το άτομο πρέπει, ο κατηγορούμενος πρέπει να απαλλαχθεί. Το αντίστοιχο στο γαλλικό δίκαιο βρίσκεται στο άρθρο 353 του ε, κώδικα ποινικής δικονομίας όπου αναφέρονται σε ε, πεποίθηση που πρέπει να έχει ε, η Επιτροπή για, την, για το ότι ο κατηγορούμενος έχει εγκληματίσει. Σε περίπτωση που η δίωξη δεν καταφέρει να αποδείξει την ενοχή, τότε πρέπει να απαλλαχθεί ο κατηγορούμενος. Να τονίσω κάτι που γενικότερα είναι γνωστό στο νομικό τομέα, ότι το αδίκημα πρέπει να ορίζει όλα τα στοιχεία του εγκλήματος, οι περιγραφές δηλαδή μιας ε, ενός βιασμού, μιας δολοφονίας δεν υπάρχουν για να ενημερώνεται το κοινό για το τι απαγορεύεται. Πρωταρχικός σκοπός είναι να ορίζουν ποια είναι τα στοιχεία του εγκλήματος, το corpus delicti που πρέπει να αποδειχθούν. Διαφορετικά έχουμε απαλλαγή του κατηγορουμένου. Το 1998 στο παλιό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθιερώθηκε μια εξαίρεση στο τεκμήριο αθότητας που πρέπει να ερμηνευτεί πολύ περιοριστικά, ειδικότερα επειδή το νέο δικαστήριο δεν την έχει ακολουθήσει σε τέτοιου είδου περιπτώσεις. Εκεί λέει, και το βλέπετε στο κόκκινο κείμενο, το ECHR το χαρακτήρισε με σχεδόν μία πορευταία τεκμήριο αθότητας επειδή δεν ήταν βέβαιο για τη γαλλική δικαιοσύνη ότι η κατοχή τέτοιες ποσότητας ναρκωτικών αποτελούσε λαθρεμπόριο. Εκεί είχαμε λοιπόν μερικό τεκμήριο ενοχής, εξαιρετική ε, περίπτωση και η αντιστροφή της, ε, του βάρους της απόδειξης ε, υπό αυτή, σε τέτοιες συνθήκες είναι αποδεκτή και, αλλά εξαιρετική. Έχουμε την πρόσθετη υπόθεση από φαντά Καταγαλίας όπου εκεί αναφέρεται το άρθρο 21.6 του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα, όπου λένε το γεγονός ότι δεν μπορεί να αιτιολογήσει κανείς του σπόρους που αντιστοιχούν στον τρόπο ζωής του ή το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να αιτιολογήσει την προέλευση ενός ε, αγαθού, περιφερειακού στοιχείου, οδηγεί στο τεκμήριο ότι το άτομο πρέπει να αποδείξει το ίδιο, φέρει το ίδιο το βαρός αποδείξεως, να αποδείξει δηλαδή την προέλευση των περιφερειακών του στοιχείων. Στο αγγλικό σύστημα του Common Law η εξαίρεση, θα, δεν θα μακρηγορήσω, η εξαίρεση για το τεκμήριο αθότητας για το βάρος της απόδειξης, συγγνώμη, γίνεται σε περιπτώσεις όπου υποβάλλει κανείς έτσι για επιστροφή φόρου και όπου τις γνώσεις της σχετικής της έχει ο εναγόμενος και εκεί η δίωξη δεν μπορεί να αποδείξει την πηγή του περιουσιακού σας Εσείς πρέπει να αποδείξετε ότι το περιουσιακό στοιχείο ε, προέρχεται από νομιμή πηγή. Φυσικά το δικαίωμα του αναγωμένου για σιωπή προέρχεται από το τεκμήριο γιατί αν δεν πει τίποτα κατά τη διαδικασία, αν παραμείνει σιωπηλός καθ' τη διάρκεια της διαδικασίας, παρόλα αυτά το βάρος των αποδείξεων το φέρει η δίωξη. Ο ενάγων. Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις που αφορούν την αυτοενοχοποίηση, το προνόμιο ε, κατά της αυτοενοχοποίησης, Γκέβγεν έναντι Γερμανίας και Γιάλοχ έναντι Γερμανίας. Αν είχαμε παραπάνω χρόνο θα μπορούσα να σας εξηγήσω περισσότερα για αυτές τις υποθέσεις αργότερα. Αλλά προς το παρόν ο χρόνος μου έχει εκπνεύσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή, πυκνή παρουσίαση όμως στηρίσατε το χρονογόρευσης. Έχετε σίγουρα δώσει με την παρουσίασή σας τροφή για πολλές απορίες. Αλλά θα τα ακούσουμε τα ερωτήματα μετά την δεύτερη παρουσίαση του κύριου Χόλγερ Μάτ που και πολύ καλά γνωρίζει το δίκαιο αλλά και τη φιλοσοφία. Συνδυάζει φιλοσοφία και δίκαιο. Είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου ποινικό Κύριε Μάτε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε και κυρία Εισηγήτρια, για το θέμα για το οποίο θα μιλήσω. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι ενώπιον σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος, Σύλλογο Σύλλογος Ποινικολόγων σας έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας, λογικά θα τις έχετε λάβει. Και αυτά που θα σας πω περιέχονται σε αυτό το έγγραφο λοιπόν. Καταρχάς πρέπει να συγχαρούμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι η πρόταση για οδηγία σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας είναι κάτι το καλοδεχούμενο. Και σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε στην παράγραφο 6, στην αρχή της παραγράφου 6, ότι σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης του τεκμηρίου αθωότητας, στόχος, ο στόχος του τεκμηρίου αθωότητας δεν μπορεί να ε, ολοκληρωθεί και δεν μπορούμε να έχουμε μια δίκαιη δίκη. Και όπως είπε και ο προλαλής σας, οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Έχουμε την ε, προφυλάκηση πριν τη δίκη, έχουμε την πρόσβαση σε δικηγόρο κτλ. Ο Ευρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος Ποινικολόγων έχει παρατηρήσει μια διάβρωση του κράτους δικαίου σε βάρος ρυθμίσεων οι οποίες ενισχύουν την εξουσία του κράτους και ταυτόχρονα μειώνουν τα δικαιώματα των υπόπτων ή των κατηγορουμένων. Και στα πλαίσια αυτά, η οδηγία αυτή για το τεκμήριο αθωότητας είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές και είναι ιδιαίτερα μεγάλη σημασίας. Κυρίες και κύριοι, το νομικό πλαίσιο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το άρθρο 82 παράγραφος 2 όπου ζητούνται ελάχιστα πρότυπα για τις ποινικέ διαδικασίες έτσι ώστε να ισχύει αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης και αυτό πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και μην ξεχνάμε βασίζεται στην εμπιστοσύνη των πολιτών της το σύμφωνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Στρασβούργου είναι καλό, δεν είναι όμως αρκετό. Δεν είναι επαρκές στην καθημερινή πρακτική των, ε, της ποινική διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αργά για τους κατηγορούμενους ή για τους υπόπτους και στο τέλος της ε, διαδικασίας υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αδυναμίες και τα μέτρα δεν επαρκούν ή δεν είναι εφαρμόσιμα. Και δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε αυτές, αυτήν την ε, δικονομική ασφάλεια. Όμως, το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο συνδέεται και με άλλα δικαιώματα. Για παράδειγμα το δικαίωμα της σιωπής ή το δικαίωμα, να, ε, το δικαίωμα μη βασανιστήριων. Το δικαίωμα της πληροφόρησης για τα δικαιώματα του υπόπτου. Ο υπόπτος πρέπει να, να καταλαβαίνει τα δικαιώματά του και να του δίνονται πληροφορίες σε γλώσσα που κατανοεί. Έχουν όμως γίνει, να το αποδεχτούμε αυτό, πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Υπάρχει σημαντική συνεισφορά, μην ξεχνάμε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επίτευξη μιας συνένεσης. Και αναφέρομαι στην τελευταία οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Δεν είναι καλή, είναι όμως ικανοποιητική. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, τον Αντωνέσκου που ήταν ο προηγούμενος εισηγητής της έκθεσης αυτής για το ότι κατάφερε να μας φέρει σε αυτή τη συνένεση. Αυτά τα δικαιώματα, κυρίε και κύριοι, και η συσχέτιση αυτών των δικαιωμάτων θα είναι αποτελεσματικά μόνο εάν λειτουργούν συμπληρωματικά, έτσι ώστε να είναι και εφαρμόσιμα νομικά, διότι διαφορετικά μιλάμε για κάτι το τελείως θεωρητικό και ουτοπικό. Τι χρειαζόμαστε δηλαδή. Χρειαζόμαστε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας και όσον αφορά τη νομική συνδρομή, ναι, πραγματικά χρειαζόμαστε μια οδηγία γι' αυτό. Και φυσικά χρειαζόμαστε και μια οδηγία για τα δικαιώματα των παιδιών στην ποινική διαδικασία. Ωστόσο, η φιλοσοφική βάση ορισμένων ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου δεν ε, αφορά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αναφέρομαι στο άρθρο 1 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αυτό το άρθρο και στις ε, οδηγίες. Το ποινικό δίκαιο βρίσκει νομιμότητα ακολουθώντας κάποιες ηθικές αξίες και κάποιες ηθικές αρχές και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι πάρα πολύ βασικό σε αυτό. Το βάρος λοιπόν των ε, αποδείξεων πρέπει να δοθεί από την κατηγορούσα αρχή. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το δικαίωμα του να μην ενοχοποιείται κανείς και το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και το δικαίωμα διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρέπει να υπάρχει η ελευθερία της ουδετερότητας η ελευθερία της ε, ουδετερότητας ε, όσον αφορά τον εξαναγκασμό συμμετοχή σε μια ποινική διαδικασία. Και αυτή είναι μια φιλοσοφική και πολιτική πτυχή η οποία λείπει από την πρόταση οδηγίας. Από το 2006, από την πράσινη χάρτα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε δει πρόοδο. Στην πράσινη χάρτα αναφερόταν ότι δεν είναι απόλυτο το δικαίωμα στη σιωπή, και αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να διαγραφεί και που πρέπει να εκλείψει με τη νέα πρόταση οδηγία. Και εδώ θα σας παραπέμψω στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα δικαιώματα του μάρτυρα στις ποινικέ διαδικασίες. Και είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να, να συμπεριληφθεί η θέση του μάρτυρα. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ στο τι γίνεται στο Συμβούλιο, γιατί αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Και αυτά που άκουσα έτσι κι αλλιώς θα τα μάθετε το Δεκέμβριο. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια τώρα. Κυρίες και κύριοι, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα πρέπει να είναι μία κεντρική αρχή εδώ. Και αυτό είναι και το ισχυρότερο επιχείρημα που έχουμε να προτάξουμε. Δηλαδή ότι όταν ο ύποπτο δεν έχει καμία ουσιαστική δυνατότητα να παραμείνει ε, ουδέτερος, παραβιάζεται το δικαίωμα της ε, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σιωπή και εμείς είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλίωση της διατύπωσης του άρθρου 6 και του άρθρου 7 παράγραφος 3 της πρότασης Οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε στοιχεία τα οποία έχουν ληφθεί μετά από παραβίαση της, των δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να μην είναι παραδεκτά. Και η διαφορά στα άλλα με τα άλλα δικονομικά δικαιώματα είναι ότι η παραβίαση του δικαιώματο τη σιωπή μετά από καταναγκασμό για παράδειγμα είναι παράλληλα και παραβίαση βασική θεμελιώδους αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και το κράτος λοιπόν δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ληφθεί μετά από παραβίαση της νομοθεσίας. Και εδώ θα σας παραπέμψω στην πρόταση πάλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι υπάρχει μία υπορήτρα στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στο άρθρο 7 παράγραφος 4, όπου λέει ότι εκτός εάν η χρήση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων δεν θα ε, αμφισβητήσει την ουδετερότητα κτλ, κτλ πρέπει να διαγραφεί διότι δεν ακολουθεί τους, τον, ε, το κράτος δικαίου. Και η πρόταση που έγινε από το Συμβούλιο στη γενική του προσέγγιση να διαγραφεί δηλαδή έτσι απλά όλη η παράγραφος είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτό. Τώρα, ολοκληρώνω λέγοντας ότι σε πολλά κράτη-μέλη ένας ε, κατηγορούμενος που αθωώνεται μπορεί να υποστεί ποινικέ ε, κυρώσεις εάν δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Αυτό δεν... Αυτό δεν ισχύει φυσικά, όπως ξέρετε, και η οδηγία δεν καλύπτει τις νομικές οντότητες. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε εσείς να ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες ή να διαβάσετε και το έγγραφο που σας έχουμε δώσει. αλλά και ο, και συνάδελφός μου, ο κύριος ε, Ζουπάντσης, μπορεί να σας μιλήσει και εκείνος περισσότερο για το βάρος της απόδειξης και της ε, αντιστροφής του. Κύριε και κύριοι, όλη η νομιμότητα του ποινικού δικαίου και της ποινική δικονομίας τίθεται υπό αμφισβήτηση εδώ και αυτό το μπέρδεμα οδηγεί σε παραβάσει σε όλο το νομικό σύστημα. Και θα ήθελα να πω τέλος ότι χρειάζεται να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των μαρτύρων σε αυτήν την οδηγία, διότι σε πολλές περιπτώσεις είμαστε άνθρωποι και είμαστε μάρτυρες σε μια κατάσταση, σε μια ποινική διαδικασία και πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα της σιωπής, το δικαίωμα της μη ενοχοποίησης σε αυτές τις περιπτώσεις. Η τελευταία πρόταση τέλος, η έκκληση που θέλω να κάνω και εγώ και ο, ποινικό, και ο δικηγορικός σύλλογος ποινικολόγων είναι να διατηρηθεί το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας που τηρήσατε τους χρόνους ομιλίας. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου και στη μέλη στην αίθουσα, Υπάρχει ένα αίτημα από τον κύριο Άλμπρεχτ. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Πριν περάσουμε στην ερώτησή του, δύο παρατηρήσεις, ερωτήσεις ίσως. Η πρώτη αφορά τους δύο καλεσμένους μας, αφορά το απαράδεκτο της ε, απόδειξης. Ξέρω ότι, όπως υπενθυμίσετε μόλις κύριε Μάτ, τα κράτη-μέλη δεν είναι ιδιαίτερα υπέρ αυτό, αλλά με αυτή την οδηγία δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς κανόνες που να αφορούν ακριβώς το μη αποδεκτό της απόδειξης. Όταν αυτή λαμβάνεται με παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ερώτημα και προς τους δυο σας. Και αφορά και τη δική μου εργασία φυσικά και των σκιωδών. Και μετά Προς εσάς κύριε Ζουπαντσίτς αναφέρατε το γνωστό διάταγμα Σαλαμπιακού, την απόφαση Σαλαμπιακού, ως μια περίπτωση ιδιαίτερως ε, εξαιρετική. Μια εξαίρεση στο τεκμήριο αθωότητας και στην αρχή του βάρους αποδείξεως που βασίζεται φυσικά στο θέμα της δίωξης. Τι θεωρείτε ότι γίνεται στο άρθρο 5 της οδηγίας όπου προβλέπεται η αντιστροφή του βάρους αποδείξεως. Βάσει της ανάλυσης σας μήπως αυτό πλήττει την ίδια την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας. Μήπως είναι αναγκαίο να ξαναδούμε αυτή την πτυχή ίσως διαγράφοντας παρέχοντας τη δυνατότητα να διαγραφεί αυτή η διάταξη. Αυτές είναι οι δυο μου Δίνω το λόγο τώρα στην αίθουσα και σας προτείνω στη συνέχεια να απαντήσετε. Έχουμε τον Γιάνν Άλμπρεχτ πρώτα απ' όλα. Έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις πολύ σημαντικές αυτές παρεμβάσεις και συστάσεις που μας δώσατε θα μας βοηθήσει στη δουλειά μας για το τεκμήριο αθότητας και την λόγω οδηγία. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ότι ξανακούσαμε πολύ ξεκάθαρο ότι στόχος είναι να προστατευτεί αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα του τεκμηρίου αθότητας μεταξύ άλλων δε και της απόλυτης προστασίας του να μην μπορεί κανείς να κατηγορεί κάποιον ε, επειδή δεν μιλάει, επειδή παρέμεινε σιωπηλός. Η σιωπή να σημαίνει δηλαδή ενοχή. Αλλά εγώ μπορεί να σιωπώ για να μην πω κάτι λάθο ή για να μην αυτοενοχοποιηθώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και αυτή η προστασία πρέπει να είναι απόλυτη. Επίσης σας συνάγω από τα συμπεράσματά σας ότι και στο πλαίσιο της νομολογίας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι σαφές αυτό. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει ένα κατώτερο επίπεδο αποδεικτικού στοιχείου που θα είναι απαραίτητο ώστε να αποδειχθεί μια κατηγορία για τις αρχές επιβολής ομοθεσίας ή για τα δικαστήρια. Δική μου εντύπωση είναι ότι φυσικά το δικαστήριο του Στρασβούργου βάζει το κατώτατο όριο, βάζει ένα κανόνα, δεν λέει όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξαίρεση στο ότι το βάρος της απόδειξης το έχει ο κατήγορος. Η κατηγορούσα αρχή. Αλλά για να, υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων πρέπει να, υπάρχει και, να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μιλάμε για αυτή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στόχος του Κοινοβουλίου ήταν και είναι όχι μόνο η εναρμόνιση ως προς το κατώτε, ε, στα ελάχιστα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά να έχουμε μια απόλυτη προστασία. Σε ό,τι αφορά την ομολογία τώρα του δικαστήριου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν υπάρχει σωστή ερμηνεία και επειδή μιλάμε για εξαιρέσεις, θα ήθελα να μας δώσετε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες για τις κατηγορίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να υπάρξουν εξαιρέσεις στο οποίο έχει το βάρος απόδειξης. Ευχαριστώ. Merci, Yann. Ε, je Ευχαριστώ Γιάννη λέει Πρόεδρος. Ε, η Μπίρκη Τσίπελ έχει τώρα το λόγο, αλλά θα σας παρακαλώ κυρία Τσίπελ να είστε, όπως ξέρετε πολύ καλά, να το κάνετε πολύ σύντομη. Θα ακούσουμε μετά μια συνάδελφο και θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών για να μπορέσουμε να έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και τις απαντήσεις και να έχουμε και χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προσπάθησα κάποτε να μάθω γαλλικά μόνη μου και ο δασκαλός μου μου είπε ότι δεν υπάρχει ούτε κανόνας ούτε εξαιρέσεις και αυτό ισχύει και για πάρα πολλούς νόμους. Κανένας νόμος δεν είναι τόσο τέλειος ώστε να ταιριάζει 100% σε όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν και καταλαβαίνω το ρόλο των δικαστών. Και ταυτόχρονα θα συμφωνήσω και με τον Γιάννη Φιλιππά Αλμπρέχτ για το ότι αν θα ήταν φρόνιμο η αντιστροφή του βάρου των αποδείξεων να αναφέρεται σε ευρωπαϊκό νόμο. Πάρα πολλές φορές έχουμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο ότι εξακολουθούμε να έχουμε αυτήν την ε, δικαστική παράδοση στα κράτη-μέλη. Δηλαδή αυτή την πολύ διαφορετική δικαστική παράδοση σε κάθε κράτος μέλος. Και εάν θέλουμε να συμπεριληφθεί αυτό στην νομοθεσία, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτήν την διαφορετική ερμηνεία και την διαφορετική χρήση της αντιστροφής του βάρους των αποδείξεων σε κάθε κράτος μέλος. Και δεν ξέρω εσείς ποια άποψη έχετε και θα ήθελα να μάθω, αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μια ενιαία νομοθεσία θα ήταν καλή. Εγώ όμως δεν πιστεύω πως αυτό είναι προς το κοινό συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λαουριστίν και να προσθέσω άλλο έναν ομιλητή, την κυρία Τσαντόφσκη. Έχετε το λόγο κυρία Λαουρέστελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου θα πάει λίγο παραπέρα. Καταλαβαίνω ότι η οδηγία αφορά καθαρά την ποινική δικονομία, αλλά αυτό που με ανησυχεί σχετίζεται με το έργο μας ε, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τις καθημερινές πρακτικές ε, όπου βλέπουμε σε όλες τις χώρες ε, ε, τις πρακτικές που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία γενικά δεν τηρούν την αρχή του τεκμηρίου αθότητας. Στην εποχή μας ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι μονοφήμες και δεν μετράει. Σε σχόλια που έχουμε στο διαδίκτυο ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημιουργούνται στοιχεία τα οποία διατηρούνται και μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή και κανείς δεν ρωτάει υπάρχει νόμιμη απόδειξη ή όχι. Μπορεί κάποιος να ενοχοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Μερικές φορές ε, οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται για χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις το εν λόγω άτομο, τα παιδιά του, η οικογένειά του έχουν καταδικαστεί από την κοινή γνώμη και αυτό μένει για πάντα. Η ερώτησή μου λοιπόν, η οδηγία αυτή περιλαμβάνει κάποια υπόνοια οτιδήποτε όσον αφορά τις πρακτικές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως και το δικαίωμα του να ξεχαστεί κανείς. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, τελευταία ερώτηση, ο κύριος Τσαντζόφσκι, Έχετε το λόγο. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω πολωνικά. Γιατί το ζήτημα είναι τέτοια σοβαρότητα που απαιτεί πολύ συγκεκριμένε και ακριβεί εξηγήσει. Για τον κύριο Μάτα θέλω να πω, η πολωνική κοινή γνώμη και η πολωνική κυβέρνηση καλωσορίζουν την πρόταση οδηγίας. Την καλωσορίζουν διότι στην πολωνική νομοθεσία ήδη έχουμε συμμορφωθεί με τις περισσότερες συστάσεις του σχεδίου οδηγίας. Και άλλωστε αυτό στηρίζει και τη δική μας ε, μακροχρόνια νομική παράδοση. Ήδη από το 15ο αιώνα ακολουθούμε ε, την αρχή στην Πολωνία ότι δεν είναι δυνατή η κράτηση και στέρηση ελευθερίας ενός ατόμου χωρίς δικαστική απόφαση. Με μόνη εξαίρεση βέβαια την κομμουνιστική εποχή. Είμαι αισιόδοξο λοιπόν. Έχω όμω και κάποιε ερωτήσει προ τον κύριο Ματ. Δύο τον αριθμό. Πρώτη ερώτηση. Είπατε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου το τεκμήριο αθότητας δεν εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Δεν είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν. Και αυτό δεν είναι μια στέρεη βάση για τις δράσεις που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι αν θα μπορούσατε να μου αναφέρετε έτσι τις πιο τρανταχτές τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν έγινε σεβαστό το τεκμήριο αθότητας στα κράτη-μέλη. Γιατί κατά την άποψή μου είναι λόγος να αναλάβουμε δράση τέτοιες περιπτώσεις. Δεύτερον, καθεστώς του μάρτυρα. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα αυτό. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει υπόψη το σύνολο των αρχών που θα πρέπει να ενσωματώνει και να εφαρμόζει ένα καλό νομικό σύστημα. Αν λοιπόν χορηγούμε στο μάρτυρα το ίδιο καθεστώς με αυτό που χορηγούμε στον κατηγορούμε, στον εναγόμενο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση κάποιων διαδικασιών, ιδίω εάν τίθεται θέμα οργανωμένου εγκλήματος. Εάν μάρτυρας και εναγόμενος έχουν την ίδια αντιμετώπιση, έχουν το ίδιο καθεστώς, ίσως το δικαστήριο να μην μπορεί να ε, λειτουργήσει. Γι' αυτό καταλαβαίνω και τις επιφυλάξεις των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τις ερωτήσεις και προτείνω να απαντήσει το καθένας, ε, να απαντήσει με το δικό του τρόπο στις 5-6 ερωτήσεις ε, στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε. Να απαντήσετε λοιπόν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τις εξαιρέσεις, για τις αρχές, για την Πολωνία και για το μη, αποδεκτό της ε, απόδειξης. Ποιος ξεκινάει. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκτός μικροφώνου κύριος ομιλητής. Έχω δύο περιπτώσεις στη Γερμανία και βγαίνει και, εναντίο, και για άλλο κατά Γερμανίας, εναντίον Γερμανίας. Στις περιπτώσεις αυτές υπήρξε παραβίαση όχι του βάρου της απόδειξης, αλλά και πίεση στον αναγόμενο να δώσει τη μαρτυρία του, δηλαδή εξαναγκάστηκε να παραβιάσει το δικαίωμά του να παραμείνει σιωπηλός. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό συνέβη με μια σχετικά έντονη πίεση επί του αναγωμένου. Και η μόνη διαδικαστική κύρωση για αυτό το μη αποδεκτό της απόδειξης ήταν ο κανόνας της εξαίρεσης. Δηλαδή, όταν πάει στο common law, ειδικότερα στο αμερικάνικο δίκαιο, αλλά και στο αγγλικό δίκαιο, έχουν κάτι το οποίο ονομάζεται exclusion tainted evidence, ε, ε, αποκλεισμό μη παραδεκτό απόδειξη, όχι μόνο απόδειξη που έχει ληφθεί μέσω παραβίαση τη αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αλλά και με αυτό που ονομάζουν φρούτα του δηλητηριώδους δένδρου. Δηλαδή αποδείξεις που προέκυψαν από παραβίαση ανθρωπίνου δικαιώματος. Με άλλα λόγια, ε, για να έχουμε ένα συνεκτικό σύστημα πενικό, θα πρέπει να έχουμε αυτό τον κανόνα αποκλεισμού όπως διαπιστώθηκε σε αυτές τις δύο υποθέσεις όπου το δικαστήριο έδωσε εντολή για αποκλεισμό των αποδείξεων που είχαν ληφθεί έτσι. Υπάρχει νομίζω και στο άρθρο 16 της συνθήκης ε, των ΗΕ κατά των βασανιστήριων κτλ. κτλ. Αν δεν ε, επιβάλλονται κυρώσεις σε τέτοιου είδους ε, παραβιάσεις, εάν δεν επηρεάζεται το αποδεκτό τους, το παραδεκτό τους, τότε δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Μπορείτε να τους περιλάβετε στο Σύνταγμα, στον κώδικα, όπου θέλετε. Να το δηλώνετε παντού. Η δεύτερη μου απάντηση θα αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν σέβονται το τεκμήριο αθεότητας. Αλλά το έχω ξαναπεί παλιότερα. Ε, προηγουμένως, συγγνώμη να το βρω μισό λεπτό. Ανέφερα προηγουμένως το Γενικό Σχόλιο 32 του άρθρου 14 της Διεθνούς Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λέει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να αποφεύγουν ειδήσει που υπονομεύουν το τεκμήριο αθότητας. Εδώ έχουμε ένα γλωσσικό πρόβλημα. Στα γαλλικά μέσα λένε «le présumé coupable», υποτιθέμενος ένοχος, που δεν σημαίνει «the presumed ο θεωρούμενος θεωρείται ένοχος, Αυτό σημαίνει. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Ακόμη και στον χώρο του διαδικτύου, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατήσουμε ουδέτερα τα μέσα. Μόλις ε, δηλώσουν κάτι και βλέπετε κάποιον με χειροπέδες ε, να τον πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα, το τεκμήριο αθωότητας ε, έχει πετάξει. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κάποια νομολογία η οποία αναφέρεται στις δηλώσεις δημοσίων αξιωματούχων τουλάχιστον που αφορούν το δεκμήριο αθωότητας του υπόπτου κατηγορουμένου. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ, άρα δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια επιχειρήματα με τον προλαλήσαντα συνάδελφο. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα γιατί χρειάζεται μια τέτοια οδηγία στον τομέα αυτό του τεκμηριωθότητας, θα ήθελα να αναφέρω σε κάτι που είπε ο νυν ε, το Μάρτιο, η κυρία Βέμπερ συγκεκριμένα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 που είναι νομική βάση ε, της συνθήκης αλλά και στο άρθρο 52 παράγραφος 3 του Χάρτη μελλοντικών Δικαιωμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί υπάρχει σαφής θέση και πρέπει να είναι και σαφής και η πολιτική θέση του Κοινοβουλίου κατ' εμέ. Η άποψη βέβαια αυτή που εκφράζω είναι η άποψη του Συλλόγου Ποινικολόγων ότι θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία από αυτή που παρέχει η νομολογία του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί αυτό είναι και ο νομικός ε, σκοπός του άρθρου 82, παράγραφος 2. Δηλαδή, να βελτιώσει την αμοιβή εμπιστοσύνη, κάτι που είναι αναγκαίο για την ε, διατήρηση της αρχής του τεκμηρίου αθότητας και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης ε, του Ευρωπαίου πολίτη στην ομολογία των άλλων κρατών, σε ό,τι αφορά τους μάρτυρες. Αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς αν θέλει να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όπως αυτή προστατεύεται στο άρθρο 1 του Χάρτη Μιλετών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέγεται ότι είναι αναπαλωτρίωτη και απαραβίαστη η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άμα θέλω να έχουμε αυτή την αρχή πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα, να προστατεύονται και οι μάρτυρες και το δικαίωμά τους να παραμένουν σιωπηλοί. Αυτή είναι η τιμή που πρέπει να καταβάλει κανείς για τέτοια προστασία. Αυτή την προστασία που παρέχει ο χάρτης ε, δυνάμει του κράτους δικαίου. Και τώρα, εν τέλει, το θέμα της χρήσης ε, των αποδείξεων που αποκτήθηκαν με παραβίαση τη νομοθεσία. Θα μπορούσε να γίνει μια διάκριση μεταξύ κάποιων δικονομικών δικαιωμάτων το οποία παραβιάστηκαν. Ειδικά όμως η παραβίαση του δικαιώματος στη σιωπή μέσω καταναγκασμού για παράδειγμα, αυτό πρέπει να οδηγήσει στην νομική επίπτωση του να μην επιτρέπεται ο δηλητηριασμένο αυτό καρπό, ο καρπός από το δηλητηριασμένο δέντρο να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο σε αποδεκτικό στοιχείο. Και στο τέλος του τριμερού διαλόγου ελπίζω να έχουμε επιτύχει, ε, δηλαδή να επιβραβευτεί επιμονή μας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ε, ευχαριστούμε για ε, όλα στις περιπτώσεις που μας παρουσιάσετε, τις προτάσεις, τις αναλύσεις σας. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά ε, όσον αφορά τα σημεία που παρουσίασαν οι συναδελφοί μου. Και τις ερωτήσεις οποίες απαντήσετε, το ζήτημα του βάρους αποδείξεως, τα όρια, οι εξαιρέσεις, το παραδεκτό ή το μη παραδεκτό των αποδείξεων, καθώς και το ζήτημα της νομολογίας και του ρόλου που διαδραματίζει και τις θέσεις μας ενδεχομένως σε σχέση με αυτήν. Εγώ θέλω να είμαστε πολύ ακριβείς και αποτελεσματικοί σε αυτό το κείμενο γιατί πρόκειται για ένα κείμενο κλειδί μαζί με τα άλλα δύο κείμενα για τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως με τα οποία αποτελεί δέσμη. Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξοι σε αυτό, την επιδίωξη των ελάχιστων επέδων να σας ευχαριστήσω λοιπόν ξανά. Θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα όσα ακούσαμε σήμερα. Πριν ε, εγκαταλείψω εδώ την έδρα, να ευχαριστήσω τον Κλοντ Μοράς για την πρότασή του να διοργανώσουμε αυτή την ακρόαση. Στιγμή κλειδί στρατηγική σημασία για αυτά τα κείμενα που εκκρεμούν ακόμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πριν διεξαχθούν οι τριμερείς διάλογοι. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ πολύ Νάταλη. Περνάμε τώρα απευθείας ε, στη τελευταία σειρά παρουσιάσεων να καλέσω τον Παύλο Τσάκη παρακαλώ να έρθει στην έδρα μαζί με τους διακεκριμένους καλεσμένους μας οι οποίοι είναι πολύ αριθμοί. Ίσως να παραδώσω και εγώ τη θέση μου όταν έρθουν πάνω. Ε, Λίμπι Μακβέι, Τζέμις Μακόλ, πρόεδρος του CCB, της e ε, Ποινικής Επιτροπής, Ιγνάτιο Πατρόνε, Ιγνάτιο Πατρόνε αναπληρωτής εισαγγελέας, ε, Ντανιέλ Κρουμπιέ, πρώην Γενικός Εισαγγελέας του Εφετίου στο Παρίσι και Ολιβιέ Τελ, επικεφαλής της Μοναδάς Δικαστικής Συνεργασίας σε ποινικά θέματα της Γενικής Διεύθυνσης δικαιοσύνη της Κομισιόν. Ε, ένα πάνελ διακεκριμένων ομιλητών. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, λοιπόν, θα κρατήσω τη θέση μου. Όχι, συγγνώμη, θα... Ζητώ συγγνώμη, συναδέλφοι, που χρειάζεται να συμπίεσουμε το χρόνο. Είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα των υπερφορτωμένων συνεδριάσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, νομικοί εδώ, επιτυχιούχοι της νομικής. Εγώ θα το συγκρίνω αυτό με τις εξετάσεις μου στο Πανεπιστήμιο και ακούσαμε και πολλά για το αγγλικό δίκαιο εδώ. Ζητώ συγγνώμη που έχουμε κάτι έτσι στριμωγμένα και να ζητήσω από τους διερμηνείς να επεκτείνουμε λίγο τη συνειδρίαση και να ευχαριστήσω όλα, να ευχαριστήσω τα μέλη που έμειναν εδώ. Το εκτιμάμε ιδιαίτερα. Εκτιμάμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε και την παρουσία σας πάλι για αυτή τη τελευταία σειρά παρουσιάσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, έχει έρθει η ώρα για το τελευταίο μας πάνελ σήμερα. Πραγματικά μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα σας ενημερώσω για τον διάλογο των πολιτών. Σήμερα το απόγευμα πιστεύω πως συζητήσαμε πολύ σημαντικά και αναγκαία πράγματα αυτές τις τρεις οδηγίες και τον οδικό χάρτη μέχρι τώρα. Έχει έρθει τώρα λοιπόν η στιγμή να τοποθετηθούμε και εμείς. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονές μας, τους πανελίστες μας. Και θα δώσω αμέσως το λόγο στην Λίμπη Μακβέη, που είναι πρόεδρος του Fair Trials International, νομικού φόρουμ για τη δίκαιη δίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κλοντ Μαρές και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που με κάλεσε. Είμαστε ένα δίκτυο με πάνω από 140 ειδικού στο ποινικό δίκαιο και το δίκτυο Fair Trials έχει συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τα τελευταία χρόνια για... και έχουμε κάνει ενημερωτικό έργο σχετικά με πολλά σημεία τη ε, δικαστική συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Πρόσφατα μάλιστα εκφράσαμε τι αντιρρήσει μα για την οδηγία για ε, τα παιδιά και θα ήθελα να σας μιλήσω για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αρχίζοντας, πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι οι διαπραγματεύσεις για αυτά τα νέα μέτρα ήταν πάρα πολύ σκληρές και η διαδικασία κατάρτισης της οδηγίας ήταν πάρα πολύ περίπλοκη. Αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε τα δικαιώματα τα οποία εσείς οι νομοθέτες τα δώσετε στα παιδιά. Υπάρχει μια περίπτωση ενός 16χρονου ο οποίος υπέστη τετράωρη ανάκριση σε ένα αστυνομικό τμήμα χωρίς δικηγόρο και χωρίς καμία στήριξη υπήρχαν δύο παιδιά από το Αφγανιστάν, τα οποία κρατήθηκαν επί δύο μήνες στη Λιθουανία σε μια φυλακή ενηλίκων. Υπάρχει ένας εκδότης εφημερίδας, ο οποίος ε, χαρακτηρίστηκε ένοχος πολύ πριν τη δίκη του στη Ρουμανία. Επίσης, υπήρξε ένας άνθρωπος που ψυχιατρική ψυχιατρική βοήθεια, δεν την έλαβε και πέρασε μήνες κράτησης, ενοχοποιώντας ο ίδιος τον εαυτό του, προτού επέμβουν οι αρχές. Και τέλος υπήρξε και η περίπτωση ενός Κινέζου υπηκό, ο οποίος ε, εκτεί ποινή 20 ετών στη Ρουμανία, μετά από μία δίκη για την οποία δεν ενημερώθηκε ποτέ. Αυτά λοιπόν που συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κρίσιμη σημασία για πάρα πολλού ανθρώπου σε όλο τον κόσμο και αυτέ οι περιπτώσει που ανέφερα είναι ένα ελάχιστο δείγμα. Πώ μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα μέτρα θα είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά και πιο στεγανά και θα παρέχουν πραγματικά προστασία στους κατηγορούμενους σε όλα τα 28 κράτη-μέλη. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε και από τις διαπραγματεύσεις και από την προσπάθεια εφαρμογής του εφιστάμενου οδικού χάρτη, τον οποίο έχουμε παρακολουθήσει πολύ στενά. Την περασμένη εβδομάδα ήρθα σε επικοινωνία για μια υπόθεση όπου ένας Ολλανδός υπήκοος κρατείται, είναι προφυλακισμένος στην Ιταλία και η διερμηνία του ε, στα γερμανικά. Όταν ζήτησε Ολλανδό διερμηνέα δεν του δόθηκε παρά τις διαμαρτυρίες εκείνου και του ε, δικηγόρου του δεν έγινε τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει. Και μετά από ένα χρόνο μετά την ε, εφαρμογή ε, της οδηγίας στην νομοθεσία και υπάρχουν ακόμα ε, προκλήσεις όσον αφορά την ε, μετάφραση και την διερμηνία για τους κατηγορούμενους. Υπάρχει και μία περίπτωση στην Πολωνία όπου ένας δικηγόρος εκπροσωπεί έναν ε, κατηγορούμενο στον οποίο ο αρμόδιος δικαστής αρνήθηκε να δώσει πρόσβαση στη δικογραφία του λέγοντας ότι εάν το κάνει αυτό θα επηρεάσει την, τις έρευνες της αστυνομίας. Και αυτό έγινε μετά την εφαρμογή της ε, αντίστοιχη ε, οδηγίας στην νομοθεσία που έγινε πέρυσι τον Ιούνιο, η οποία προβλέπει να παρέχονται πληροφορίες χωρίς καμία παρέκκληση, χωρίς καμία εξαίρεση. Οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν να αρνούνται να εφαρμόσουν την αυτή. Παρά λοιπόν το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η νομοθεσία, στο χαρτί και ισχύει, εξακολουθούν να ε, υπάρχουν εμπόδια και να μην απολαμβάνουν οι τα δικαιώματα που πρέπει. Έχουμε λάβει λοιπόν εμεί πληροφορίες για αυτές τις τρεις ε, οδηγίες, για αυτές τις τρεις προτάσεις, όμως πιστεύω ότι τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από την εφαρμογή των δύο πρώτων οδηγιών θα ε, βοηθήσουν πάρα πολύ τις επόμενες. Πρώτο ζήτημα, το θέμα της ε, Πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή προκύπτουν από την έλλειψη ξεκάθαρης καθοδήγησης και ε, διατύπωσης των δύο πρώτων οδηγιών. Έχουν ε, μείνει πάρα πολλές, ε, ε δυνα, δυνατότητες ερμηνείας στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη θα αναγκαστούν να κάνουν συμβιβασμού στην ερμηνεία των οδηγιών. Υπήρξε και μία ε, συζήτηση στο Λονδίνο πριν από δύο εβδομάδες όπου συζητήθηκε το ότι οι συμβιβασμοί μπορούν μεν να δώσουν μια βραχυπρόθεσμη λύση, όμως αναγκαστικά κάποια στιγμή θα κληθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί. Και αυτό σίγουρα δεν θα ευχαριστήσει όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, επίσης ε, αντίστοιχα προβλήματα στο, στην οδηγία για την προστασία των παιδιών. Εμείς έχουμε επισημάνει ορισμένες ελλείψεις. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις εξατομικευμένες αξιολογήσεις ανηλίκων και όσον αφορά την μετατόπιση του βάρους ε, της απόδειξης. Κάτι που ακούσαμε πριν από λίγο. Ελπίζουμε πως η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα λάβει υπόψη τις παγίδες που περιέχουν οι συμβιβασμοί και θα προσέξει τη διατύπωση. Έπειτα, όσον αφορά την επιβολή. Οι πρώτοι δύο δικοί χάρτες ε, αντιμετώπισαν προβλήματα στην εφαρμογή εξαιτίας των ελλείψεων συγκεκριμένων διατάξεων για τις ε, παραβιάσεις των ε, διατάξεων και έγιναν αναφορές μόνο στις υποχρεώσεις των κρατών μελών να δώσουν σε ε, και κατηγορούμενους το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τις αρχές και το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε διάφορες διασφαλίσεις. Αλλά δεν υπήρχε καμία καθοδήγηση σε ποια ένδικα, ε, όσον αφορά τα ποια ένδικα μέσα θα έχουν στη διάθεσή τους. Επίσης, υπάρχει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όμως αυτή παραμένει ε, ανεφάρμοστη. Η πρότασή μας περιέχει ορισμένες ε, διατάξεις σχετικά σχετικά με τα ένδικα μέσα. Όμως η πρόταση οδηγίας δεν παρέχει καμία ε, τέτοια διαταξή ού, ούτε για την οδηγία για τα παιδιά, ούτε για την δεύτερη οδηγία. Έπειτα, υπάρχει το θέμα της διασύνδεσης και της συνέπειας, όπου ανέφερε και ο καθηγητής Πομπκίνλε νωρίτερα. Σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο, ο νομοθέτης πρέπει να λάβει υπόψη του τη διασύνδεση. Ο δικός χάρτης καθιστά σαφές ότι σε αυτήν την βήμα προς βήμα προσέγγιση στην νομοθεσία χρειάζεται συνολική συνέπεια και πρέπει να διασφαλιστεί αυτή, διότι υπάρχουν προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των τριών πρώτων οδηγίων και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους κατηγορούμενους ή για τους υπόπτους, ε, υπόπτους να ε, απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους χωρίς να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο που αναφέρει τρίτη οδηγία, η οποία δεν θα εφαρμοστεί για τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης, υπάρχει και η ανάγκη ε, συνοχής ανάμεσα στις οδηγίες και αυτό απειλείται από τις τρεις νέες προτάσεις. Η πρόταση οδηγίας για νομική συνδρομή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που καλύπτει η οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο και αυτό το ακούσαμε ήδη πάρα πολλές φορές σήμερα. Έπειτα, το Συμβούλιο πρότεινε για το άρθρο 6α ορισμένες αλλαγές, ορισμένες τροποποίησεις για, το, για την οδηγία για τα παιδιά. Όμως δεν υπάρχει κανένας παραλληλισμός, καμία ομοιότητα με την οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Αυτό λοιπόν που μας οδηγεί στο ότι τα παιδιά θα έχουν ακόμα λιγότερη προστασία από ό,τι πριν. Ελπίζουμε λοιπόν η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να θέσει προτεραιότητες όσον αφορά το πακέτο δικονομικών δικαιωμάτων στην ε, σύνταξη των μέτρων. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική η κατάρτιση, η ποινική κατάρτιση. Δυστυχώς δεν υπάρχει αναφορά στην κατάρτιση των ε, αρμόδιων και έχουμε τονίσει το πόσο σημαντικό είναι αυτό επανειλημμένα. Η οδηγία για τα παιδιά ε, περιέχει μέτρα κατάρτισης και μέτρα μάλιστα κατάρτισης των συνηγόρων υπεράσπισης, κάτι το οποίο χαιρετίζουμε. Δυστυχώς όμως ε, δεν υπάρχει ούτε στην ε, οδηγία για νομική συνδρομή, ούτε για την οδηγία των τεκμηριωθότητας κάποια τέτοια διάταξη. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ακόμα περισσότερη δράση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τα δικονομικά δικαιώματα. Η προφυλάκηση έχει ήδη επισημανθεί ως ένας νευραλγικός τομέας και χρειάζεται η ανάγκη νομοθεσίας, εφαρμόσιμης νομοθεσίας για τους υπόπτους και τους κατηγορούμενους. Και επίσης να μην ξεχνάμε το ζήτημα των οπτικοακουστικών ε, μέσων, της, ε, των ηχογραφήσεων και μαγνητοσκοπήσεων και αυτό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι όλου του πακέτου μέτρων για τα δικονομικά δικαιώματα και όπως είπα και πριν πρέπει πραγματικά να ε, δούμε το ζήτημα των ενδικών μέσων διότι διαφορετικά δεν θα μπορούν να τα ε, απολαμβάνουν οι κατηγορούμενοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλότερο τον κύριο Τζέμις Μαγγέλ, πρόεδρο της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου της ΕΣΥΜΠΗ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που προσκάλεσε το CCB σήμερα για να πούμε και εμείς την άποψή μας. Και βέβαια εγώ πρέπει να πω ότι η Επιτροπή σας έχει κάνει πολλή δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά και αυτό δεν διαφεύγει της προσοχής μας και πρέπει να σας πω ότι είμαστε ανακουφισμένοι που η Κομισιόν και η Επιτροπή σας ε, εξετάζει αυτά τα ε, μέτρα, γιατί αυτό το μέτρο που πρότεινε το Συμβούλιο, το μέτρο C, θα παραβίαζε πολλές διατάξεις και θα είχε μεγάλη ζημία αυτό για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη και γι' αυτό εκ μέρους όλων των ε, δικηγόρων θέλω να σας ευχαριστήσω. Και να πω καταρχάς ότι συμφωνώ με ό,τι είπαν ε, ιδίως οι Λίμποι και ο Χόλγκερ. Ο μεγάλος ε, εχθρός, ε, στην Άσο και ο κύριος Ντένις Ντεγιόγκ είναι ότι πρέπει να πάρουμε μία θέση καταρχήν. Τα οικονομικά επιχείρηματα λοιπόν είναι ο μεγάλος εχθρός αυτή την αίθουσα. Και το ακούμε από διάφορους σχολιαστές και από το Συμβούλιο. Εμείς οι δικηγόροι υπεράσπισης τα έχουμε ξαναδεί. Το έργο το έχουμε δει πολλέ φορές. Όταν ε, εισήχθησαν ε, αυτές οι διατάξει ε, για τα εντάλματα σύλληψη. θέλαμε να μπουν ασφαλιστικέ δικλείδε για να υπάρξουν κάποια αντίβαρα. 12 χρόνια μετά δεν έχει γίνει αυτό. Και μιλάμε για τον Ευρωπαίο κατήγορο. Πώς θα δώσετε περισσότερες εξουσίες αν δεν υπάρχουν αντίβαρα. Υπάρχουν κάποιοι που πείθονται από τα οικονομικά επιχειρήματα. Οπότε θέλω να σα δώσω ένα σύντομο παράδειγμα μια υπόθεση με ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη και για να σα εξηγήσω γιατί κάθε δικηγόρο και κάθε βουλευτή πρέπει να καταλάβει ότι θα επηρεαστούν αρνητικά για τη μηγορία των δικαστηρίων. Ε, μιλάμε για αυτούς που δεν έχουν μέσα για να ε, βρουν δικόρη περάσπιση και να τον πληρώσουν. Συλλαμβάνεται ένας ε, πελάτης στην Ιρλανδία και πρέπει να δικαστεί στη Φραγκφούρτη. Τι κάνω εγώ ως δικηγόρος υπεράσπιση. Αν με πληρώσει θα τηλεφωνήσω στον καθηγητή ΜΑΤ, θα μιλήσω εδώ με τις γερμανικές αρχές. Έτσι γίνεται σε πολλές περιπτώσεις που επιλύονται χωρίς να απαιτηθεί κάθυρξη. Και κάποια νομικά συστήματα πολλές φορές λαμβάνω υπόψη ε, την καλή διαγωγή, καλή πρώτερη διαγωγή. Σε άλλες περιπτώσεις όμως δεν λαμβάνεται αυτό υπόψη. Εάν τώρα εγώ ε, δεν λαμβάνω αμοιβή, δεν μπορώ να κάνω αυτά τα τηλεφωνήματα για αυτή την πολύ λογική αντιμετώπιση της ε, υπόθεσης. Αν λοιπόν δεν έχει πρόσβαση ε, σε δικηγόρο το άτομο, Και μάλιστα είναι πολύ δυσανάλογες. Πολλές φορές οι που επιβάλλονται ε, γεμίζουν οι φυλακές με άτομα που κλέψανε ε, κότες. Για παράδειγμα. Πρέπει να μπει, ε, πρέπει να γίνει μια δοκιμή αναλογικότητας. Αυτός που δεν έχει χρήματα λοιπόν, τι παθαίνει, συλλαμβάνεται, προφυλακίζεται, σίγουρα, λαμβάνει περισσότερο χρόνο η εκδίκαση υπόθεσης, Ο άτυχος άνθρωπος αυτός θα παραμείνει σε προσωρινή κράτηση για πολύ, ε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να του οριστεί δικηγόρος. Και ο καταλογισμός, ο υπολογισμός γίνεται στο τέλος γιατί να μην γίνει στην αρχή. Γιατί το ανθρώπου αυτού έχει διαταραχθεί και η οικογενειακή του ζωή, έχει μείνει προφυλακισμένος και υπάρχει και τεράστιο ε, άχθος για τα δικαστήρια με υποθέσεις που κρατάνε τόσο καιρό μέχρι να εκδικαστούν. Πρέπει να γίνει επιτέλους ε, η πρόταση και θα ήταν ντροπή να περάσει το Συμβουλίο στην προκειμένη περίπτωση. Στηρίζουμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Πρέπει να ενισχυθεί. Κατακλείδη από τους δικηγόρους υπεράσπισης Έχουμε εμπειρία, καθημερινή εμπειρία. Γιατί αυτά που προτείνουν οι κυβερνήσεις ε, ε, ουσιαστικά καταστρέφουν την εμπιστοσύνη. Οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς. Πρέπει λοιπόν να τους αναγκάσετε αυτοί να σας πούν ε, που προωθούν αυτά τα οικονομικά επιχειρήματα τι θετικό φέρουν. Και έπειτα να σας μιλήσω για το κόστος, το τεράστιο και των εφέσεων όταν κάποιος δεν έχει εκπροσωπηθεί σε πρώτο βαθμό. Δεν είναι αυτά τα οικονομικά επιχειρήματα ευσταθή. Και δύο-τρία άλλα σχόλια. Δεν σας ενθαρρύνουμε απλά και μόνο να κάνετε προτάσεις για μέτρα, για να κάνετε προτάσεις για μέτρα, αν δεν βελτιώσουν την κατάσταση δεν χρειάζεται καν. Και συμφωνώ αυτό που είπε ο καθηγητής Ματ. Δεν είναι αποτελεσματική η προστασία του Στρασβούργου για τους πελάτες μας σε καθημερινή βάση. Θέλουμε κωδικοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και βελτίωση των πρακτικών. Είναι αργά το βράδυ, δεν έχω να πω και πολλά περισσότερα, τα έχουν πει ε, οι προλαλήσαντες και τα έχουμε γράψει και σε διάφορα έγγραφα τοποθέτησης. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαγγίλ. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ινιάτσιο Πατρόνε, αναπληρωτή εισαγγελέα του Ανωτατού Δικαστηρίου, Παρακαλώ κύριε Πατρόνε. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μερικοί από σας θα εκπλαγούν ίσως που είμαι ο πρώτος εγγελέας που μιλάει σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα και ουσιαστικά συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Είμαι πεπισμένος προσωπικά Ίσως να είμαι Ιταλός, αλλά ακολουθώ τον Μπεκαρία που αναφέρθηκε. Αλλά το αναφέρω αυτό και από πρακτική άποψη, την οποία θα σας περιγράψω αμέσως τώρα. Ο μηχανισμός αμοιβέ αναγνώρισης η κυρία βουλευτής, ε, δεν θυμάμαι το όνομά της, ζητώ συγγνώμη, παρενέβη στην προηγούμενη συζήτηση, ανέφερε το γεγονός ότι, ότι ανέφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έννοια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ήταν κάτι κουραστικό. Φανταστείτε τι κούραση έχω εγώ που κάνω τη δουλειά αυτή εδώ και 33 χρόνια και που από το 99 μόλις είδα να προτείνεται κάτι τέτοιο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν είχε ασχοληθεί. Εκείνη την εποχή αποτέλεσε στοίχημα, σίγουρα βασισμένο σε σημαντικά στοιχεία αλλά μεροληπτικά στην κοινή συμμετοχή στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Κάποια, λοιπόν, κάποιος ισχυρισμός ε, διαφύλαξης των μεγάλων αρχών και κάποια ανάγκη αντιμετώπισης ε, εγκληματικότητας που γινόταν όλο και πιο διακρατική. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρξε ένα πρώτο κύμα διατάξεων και μέτρων που ξεκίνησαν από το 2001 μέσα σε μια μανία να υποστηρίξουμε την ασφάλεια. Ελάχιστη προσοχή δώσαμε τότε στη θέματα της υπεράσπασης και αυτή η ελάχιστη προσοχή οδηγεί σήμερα στο ότι με τη συνθήκη με τη συνθήκη της Λισαβόνα όπου έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες με αποτέλεσμα να γίνουν ελπίζουμε πιο αποτελεσματικέ, Εδώ έχουμε πλέον την απόλυτη αναγκαιότητα να ενοποιήσουμε το πλαίσιο των δικαιωμάτων υπεράσπιση. Είναι απολύτω αναγκαίο διότι διαφορετικά υπονομεύεται η εμπιστοσύνη, όχι αυτή που βρίσκεται στα χάρτια, η πραγματική εμπιστοσύνη των πολιτών μας που είναι το μόνο δημοκρατικό θεμέλιο πάνω στο οποίο σε ένα μη ομοσπονδιακό σύστημα και που όπως έχουν σήμερα τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνει ομοσπονδιακό θα έχει διατάξεις που ισχύουν σε όλες τις χώρες. Εγώ προσωπικά λοιπόν όχι απλά χαίρομαι που εγκρίθηκαν οι τρεις οδηγίες που ισχύουν ήδη είμαι υπερευτυχής ή μάλλον θα ήμουν υπερευτυχής αν μπορούσαμε να εγκρίνουμε γρήγορα και τις τρεις οδηγίες που συζητήθηκαν σήμερα. Ειδικότερα αυτήν ε, που συζητήσαμε αργότερα, αλλά που κατά κάποιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο απόψη αρχής αποτελεί το θεμέλιο για όλο τον υπόλοιπο τομέα. Η οδηγία για το δεχμήριο αυτό που φοβάμαι εγώ είναι ότι αν δεν καταλήξουμε σε κάποιο καθορισμένο πλαίσιο προστασίας, το οποίο να εναρμονίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα δικαιώματα των μερών μιας ποινική διαδικασίας, η έλλειψη εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμα θα υπονομεύσει την νομιμότητά του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ότι θα βοηθήσει την εγκληματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι το ποινικό σύστημα πρέπει με τις μέγιστες εγγυήσεις να αποδίδει κιόλα ε, φαίνοντας αποτελέσματα υπερασπιζόμενο το κοινό καλό. Είναι μια ισορροπία που πάντα υπήρξε μεταξύ των δικαιωμάτων του ατόμου και του δικαιωμάτων της κοινωνίας να τιμωρεί τα δικήματα. Είναι δύσκολη η ισορροπία, αλλά απολύτως απαραίτητη. Ο χώρος ε, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν πρέπει να ευνοεί την ατιμορρησία. Δεν μπορούμε να αποφεύγουμε τις ευθύνες μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να μην επιτρέπει να περνάμε τα σύνορα να αλλάζουν τα δικαιώματά μας. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει στις αρχές να συλλέγουν τα αποδεικτικά στοιχεία όπου θέλουν, με το μέσο που θέλουν και κυρίως χωρίς να υπάρχει εγγύηση ενός ελάχιστου στάνταρ. Εδώ ξεκινάω το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας μου. Διότι ε, ανέφερε ο εισαγγελέας Σάρφστον πρόσφατα ένα ζήτημα ε, σε μια ομιλία του πολύ ενδιαφέρουσα, την υπόθεση ΕΜΕ δεν θέλησε να κατονομαστεί το πρόσωπο αφορούσε ένα, μια υπόθεση μεταξύ Ιταλίας και Βελγίου. Ο Γενικό Εγγελέα Άπστον, που δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά θαυμάζω για την ακριβιά του, στο τέλο είπε ότι κοιτάξτε, χρόνο για να ορίσουμε πρότυπα περί ποινική ε, δικαιοδοσίας ε, χρειαζόμαστε. Όσον αφορά τις αστικές διαφορές, έχουμε πλήρη νομοθεσία που λειτουργεί. Είναι ενδιαφέρουσα ένα σύστημα το οποίο κατανέμει πολύ σωστά τη δικαιοδοσία. Βέβαια, το αστικό δίκαιο αφορά τους ιδιώτες. Αν δεχτώ εγώ να έρθω στο Βέλγιο αντί για την Ιταλία, στο ποινικό δίκαιο τίθεται το εξή ερώτημα. Υπάρχουν σημαντικές αποφασιστικές ε, συνέπειες. Ποιος είναι αρμόδιος λοιπόν, το ποιος είναι αρμόδιος ορίζει το δίκαιο που θα διέπει την πράξη και τη διαδικασία. Το δίκαιο αυτό ως κυρίαρχο δίκαιο. Δεύτερον, αποτρέπει τον κίνδυνο να υπάρχουν ταυτόχρονα δύο έρευνες ή περισσότερες έρευνες για την ίδια υπόθεση γιατί για τα διασυνοριακά εγκλήματα. Είναι σχεδόν φυσιολογικό πια να γίνονται έρευνες πολλαπλές ε, σε τρεις-τέσσερις χώρες. Και αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε. Και ο κύριος Αρστόν λέει ακριβώς αυτό. Δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί σε μεταγενέστερη φάση αφού κάποιος έχει καταδικαστεί και απαλλαχθεί σε μια χώρα. Χρειάζεται ένας ε, μηχανισμός πολύ γρήγορου ορισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πλαίσιο των οδηγιών θα πρέπει να εγκριθεί και σε αυτό πρέπει να προσθεθεί μια, ε, ένα σύστημα κατανομής της αρμοδιότητας μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο τέταρτος εμπειρογνώμονας στο πάνελ μας σήμερα είναι ο Ντανιέλ Λεκρουμπιέν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν και έξι χρόνια εδώ στη μόνιμα αντιπροσωπεία ε, της Γαλλίας. Ε, άρχισα μετά από το Τάμπερε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τότε υπήρχε μεγάλη δυναμική Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια πιο σωροπημένη απάντηση στα ερωτήματα. Από το 2004 και μετά κάπως ε, αποδυναμώνεται η δυναμική και έχουμε την απόφαση πλαίσιο για τα δικονομικά δικαιώματα. Το δείχνει αυτό η τότε απόφαση. Πρέπει να σας πω ότι με την πρόταση εκείνη υπερβαίναμε την αρχαία αμοιβαία αναγνώριση που ήταν η βασική αρχή μέχρι τότε και αυτό για λόγους ευκολίας. Στόχος ήταν όμως να έχουμε τουλάχιστον κάποια κοινά πρότυπα και προσεγγίζοντας τον πυρήνα του δικαστικού συστήματος κάθε, χρόνο, ε, κάθε χώρας ήταν πολύ λεπτό το θέμα και γι' αυτό χρειάστηκε να περιμένουμε τη Σουηδική Προεδρία το 2009 Οπότε και καταρτίστηκε ο δικός χάρτης ε, βάσει το οποίο εργαζόμαστε σήμερα. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η συνεδρία. Πέντε χρόνια χρειάστηκαν για να έχουμε δικό χάρτη για, τα δικονομικά, ε, για τις δικονομικές εγγύησεις από το Συμβούλιο. Και πέντε χρόνια χρειάστηκαν για να γίνουν αυτά που έγιναν μέχρι τώρα. Τι χρειάζεται, θα περιμένουμε άλλα πέντε χρόνια τώρα ή τι θα γίνει στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν θέλω να τι είπαν οι προλαλήσαντες, γιατί θέλω να πω ότι συμφωνώ και με τους συναδέλφους και απριόρι συμφωνώ και με όλες τις προτάσεις που διατύπωσαν. Σε ό,τι αφορά την ε, ε, νομοθεσία περί ε, ευεργετήματος παινίας είναι το βασικό ζήτημα για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Είναι θεμελιώδης δικαίωμα, αλλιώς θα είναι και όλα τα άλλα δικαιώματα απλά τυπικά και όχι Και θα έλεγα ότι πρέπει να πάμε και πολύ πιο μακριά. Και για τους ανηλίκους αλλά και για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολία θα έπρεπε να έχουμε συστηματικοποιημένη ε, ε, αρχή ε, δωρεάν παροχή του ευεργετήματος παινίας. Κάθε ανήλικος θα έπρεπε να έχει την στήριξη ενός δικηγόρου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Για το άρθρο 7 συγκεκριμένα τώρα, τις οδηγίες για τους ανηλίκους, και για τα θύματα εμπορίας προσώπων. Νομίζω ότι αυτό με το σημείο 32 πράγματι είναι ασαφές και πρέπει να διευκρινιστεί. Θα επανέλθω. Φυσικά μπορεί να τεθεί το ερώτημα αυτή η δημιουργία του χώρου δικαιοσύνη, ασφάλεια ελευθερία. μπορεί στα δικονομικά συστήματα να περιοριστεί στην πρόταση που είχε γίνει πριν 5 για να μην πω πριν 10 χρόνια τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να έχουμε μια νέα πρόταση από την Κομισιόν. Ίσως καλό θα ήταν αυτός ο δικός χάρτης ε, να επικοιμηνθεί σε κάποιους άξονες, όπως υπόθηκε παραδείγματος χάρη για τους εφαρμοστέους κανόνες ό,τι αφορά την προσωρινή κράτηση ή τους όρους κράτησης ή το μητρό για τους ε, αλλοδαπούς, το ποινικό μητρό. Πάντως πρέπει να είμαστε ε, λογικοί δεν είναι κατά ανάγκη και το καλύτερο δυνατό να νομοθετούμε συνεχώ με νέα κείμενα. Για τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι το σημαντικό είναι πραγματικά να εφαρμοστεί η οδηγία ε, την οποία συζητούμε. Για να έχουμε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό νομικό κόρπους. Πρέπει να δώσουμε πνοή, να δώσουμε ζωή σε όλες αυτές τις διατάξεις. Και η Κομισιόν θα πρέπει να ασκεί ρόλο ε, ελεγκτή, ελεγκτικό ρόλο για την εφαρμογή αυτή τη οδηγία από 1 Δεκεμβρίου και μετά. Και να βασιστεί βέβαια και στου επαγγελματίε του κλάδου, Επενδύοντα στην εκπαίδευση, επενδύοντα στις αξιολογήσει των ε, δικαστικών συστημάτων, ώστε για αυτά τα κατώτατα πρότυπα και κανόνε να έχουμε πραγματικά ε, εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο κατώτατο αυτό επίπεδο. Και για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. η ένταξη, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα αποφασιστικό βήμα. Και ένα θέμα που μπορεί να σας φαίνεται ελάσσονο σημασίας, αλλά για μένα είναι σημαντικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι από την 1η Δεκεμβρίου ο τομέας τη δικαστική συνεργασίας ε, στο, στα θέματα ποινικού δικαίου θα υπάγεται ε, σε ένα κοινό πλαίσιο. Θα πρέπει να ορίσουμε στρατηγικέ σε θέματα ποινική δικαιοσύνη. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς τα έμπρο για την πραγματική προστασία των δικαιώματων που συζητούμε. Θα σα δώσω ένα δύσκολο παράδειγμα πολύ δύσκολο παράδειγμα, για να προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι εννοώ. για την νεανική παραβατικότητα και συγκεκριμένα παιδιών από οικογένειες Ρωμά η κυκλοφορία, η ελευθερία κυκλοφορίας έχει αυξήσει και πολύ σημαντικά μάλιστα αυτή την παραβατικότητα από παιδιά Ρωμά. Μπορούμε να πούμε πολλαπλά το λύνουμε καταργώντας αυτή την ελευθερία κυκλοφορίας, ε, επαναπροωθώντας ε, τα παιδιά στις χώρες τους, ε, ας, στείλουμε πίσω τους Ρωμά στις χώρες τους στην εξαθλίωση. Φυσικά και δεν είναι αυτή η δική μου άποψη, δεν είναι αυτή η λύση. Ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οικονομικές απαντήσεις δίνει, χρηματοοικονομικές. Αρκεί αυτό όμως. Έχουμε να δώσουμε απαντήσεις απέναντι σε αυτό το πρόβλημα της παραβατικότητας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν μου πει κάποιος ότι ναι, ε, θα ικανοποιηθώ πάρα πολύ που να απάντηση αυτή, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Στο Παρίσι, σεβόμαστε όλους αυτούς τους κανόνες για τους οποίους έγινε λόγος. Παρ' όλα αυτά, ε, κρατούνται ε, μπαίνουν στα κρατητήρια παιδιά πάνω από 13 ετών. Ένα τρίτο των ανήλικων παραβατών είναι κάτω από 13. Τι τους κάνουμε αυτούς? Τους ξαναβγάζουμε αυτούς τους νέους στο δρόμο, αυτά τα παιδιά. Και δεν ξέρουμε ούτε το όνομά τους, ούτε που μένουν, ούτε ποιος έχει την επιμελιά τους, ποιος τους συνοδεύει. Αυτή είναι η απάντηση που δίνουμε ως Ευρώπη. Αυτή είναι η απάντηση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, της γαλλικής δικαιοσύνης. Εγώ ως και εισαγγελέα ε, στο εφετείο του Παρισιού. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι, δεν το κρύβω. Που έχουμε αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουμε ποια είναι ουσιαστικά. Και τα πετάμε ε, στο δρόμο και ουσιαστικά τα ρίχνουμε στα χέρια αυτών των ε, κυκλωμάτων εμπορίας που τα εκμεταλλεύονται. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Δύο είναι ουσιαστικά οι απαντήσεις. Η μία είναι να επιτεθούμε σε αυτά τα κυκλώματα και η δεύτερη απάντηση βέβαια να προστατεύσουμε τους ανηλίκους αυτούς. Στην πρώτη ε, περίπτωση, πώς επιτιθέμεθα σε αυτά τα κυκλώματα. Και η Ρουμανική αστυνομία έχει κάνει πολλά. Τι έγινε όμως, φεύγουν από το Παρίσι αυτά τα παιδιά, αλλά δεν ξέρουν που πάνε μετά. Δηλαδή δεν υπάρχει μια παρακολούθηση, μια συνέχεια στο, στην ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων. Τι γίνεται, μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεύτερος άξονας, προστασία των ανηλίκων. Να τα συνοδεύουμε, τα παρακολουθούμε κατά κάποιο τρόπο. Μεγάλες αρχές, αλλά είναι και, υπάρχουν και περιορισμοί. Γιατί υπάρχει και διάσταση δικαίων. Το είπαμε, πρέπει να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες και εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί είναι η δυσκολία. Και ακριβώς εκεί έγκυται η όλη προσπάθεια. Πρέπει να ορίσουμε στρατηγικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το Κοινοβούλιο είναι στην τέλεια θέση. Έχετε την νομιμοποίηση, την ευρωπαϊκή νομιμοποίηση. Εκλέγεστε από τους πολίτες. Έχετε ε, αυτή την ε, αξία ε, την προστατευτική. Γι' αυτό θα πρέπει να καθορίσετε τις στρατηγικές για να δώσετε πραγματικές απαντήσεις στην ποινική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεκριβιέ. Ας περάσουμε στον κύριο Τέλ. Έχετε λίγα λεπτά. Εκπρόσωπος του Γενικής Διεθνής Δικαιοσύνης στον τομέα του ποινικού δικαίου. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας από το 2009 με τη συνθήκη της Λισαβόνας και την κοινοτική μέθοδο που εμπλέκει το Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον οδικό χάρτη του 2009 πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές πρόοδους όσον αφορά το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της ενίσχυσης των δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών και στο δικαίωμα ισότιμης δίκης Έχουμε πολλές προκλήσεις ακόμα. Πρώτα απ' όλα η υλοποίηση. Δεν είναι και το πιο απλό. Όπως ξέρετε, υιοθετήσαμε τρεις οδηγίες, μετάφραση διερμηνία, δικαίωμα ενημέρωση, δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο μεταφορά τους, η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο. Και εγώ το γνώριζω καλά. Θα θίγει σημαντικές προκλήσεις δικαστικές, ε, επιχειρησιακές ε, και ε, δικαστικές. Η Κομισιόν εργάζεται ταχαίως για την ενσωμάτωση αυτών των ειδικιών στα κράτη-μέλη. Έχουν ήδη παρέλθει οι προθεσμίες ενσωμάτωσης για δύο από αυτές και η Κομισιόν αξιολογεί τακτικά την ποιότητα της ενσωμάτωσης στα κράτη-μέλη. Δύο παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα. Αυτές οι οδηγίες σε ορισμένες διατάξεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από τους αναγόμενους ως ασαφής δικαίωμα, ως ε, δικαίωμα σε διερμηνία για παράδειγμα. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν οι προκλήσεις ε, οργανωτικής φύσης, η δημιουργία ε, ομάδων ε, διερμηνέων μεταφραστών, η πρόσβαση στην δικογραφία, σε ποιο στάδιο της έρευνας, κρίσιμο σημείο στην ενσωμάτωση της οδηγίας ε, για το δικαίωμα ενημέρωσης και μετά υπάρχουν και δικαστικές προκλήσεις. Η οδηγία για τη διερμηνία αναφέρει τη μεταφράση των ουσιοδών εγγράφων. Ποια έγγραφα είναι τα ουσιοδή Η διαπραγμάτευση αυτών των οδηγιών οδήγησε σε ασαφείς έννοιες που οδηγούν σε ερμηνείε, οι οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρουν ανάλογα με το κρατούμενο μέλος. Δεύτερον, πρέπει να ολοκληρώσουμε το οικοδομά με την υιοθέτηση των τριών οδηγιών που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα που παρουσιάστηκαν από την Κομισιόν τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτές οι οδηγίες ενισχύουν το τεκμήριο αθεότητας, την προστασία των ανηλίκων, και την καθιέρωση προσωρινή νομική συνδρομή για τα άτομα που του έχει στερηθεί η ελευθερία του. Αυτό συμπληρώνεται από δύο συστάσει τη Κομισιόν για τα ευάλωτα άτομα και τη δικαστική αρρωγή και τα κριτήρια επιλεξιματικότητα. Οι επιπτώσει στα εθνικά δίκαια θα αξιολογηθούν από την Κομισιόν σε δύο χρόνια. Είναι προφανέ ότι η ενσωμάτωση αυτών των δικαιών αποτελεί βάρο και επηρεάζει τη διαπραγμάτευση των νέων προτάσεων. Το βλέπουμε πολύ καλά. Δύο λόγια τώρα για κάθε μία από τις οδηγίες. Η οδηγία για τα παιδιά είναι η πιο μεγάλη και πιο σημαντική κατά την άποψή μας. Είναι ουσιώδης σημασία διότι αφορά όλα τα δικαιώματα ε, μιας κατηγορίας ε, ατόμων, των παιδιών, κατηγορία που εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική δικαιοσύνη προσαρμοσμένη στα παιδιά. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τα παιδιά στι δικονομικέ διαδικασίε. Επιβάλλεται λοιπόν πολιτικά να τους διασφαλίζουμε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας στη στην ε, ποινική δικονομία. Για μας το σημαντικότερο είναι το δικαίωμα υποστήριξη από δικηγόρο. Δεν πρέπει να το αποδυναμώσουμε. Η αρχή είναι απλή. Κάθε παιδί όταν το, για διάπραξη ενός εγκλήματος πρέπει να λαμβάνει την υποστήριξη ενός δικηγόρου όταν ανακρίνεται από την αστυνομία. Αυτό που ισχύει είναι η προσωπικότητά του, το παρελθόν του, το ποινικό του μητρό, οι δυνατότητες επανενταξής του και όλα αυτά θα επηρεάσουν τη σοβαρότητα της κύρωσης, της ποινής. Η οδηγία που αφορά το τεκμήριο είναι μια καινοτομία από νομοθετική άποψη. Χωρίς την τήρησή της, τα δικονομικά δικαιώματα και τα υπόλοιπα δικαιώματα δεν είναι παραπλάνες. Τι να κάνει κανείς ένα δικηγόρο αν κανείς ε, δεν σέβεται το δικαίωμά σας να μην αυτό ενοχοποιηθείτε. Το τεκμήριο αθεότητας φυσικά υπάρχει σε πολλά δικαστικά συστήματα, αλλά η εφαρμογή του πρακτικά δημιουργεί προβλήματα. Δείτε τις διάφορες αποφάσεις του δικαστήριου του Στρασβούργου που αμφισβητούν πολλές πρακτικές σε κράτη-μέλη. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά σήμερα υπάρχει συνένεση μεταξύ των κρατών μελών στο ότι χρειάζεται για να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο σύνολο κοινών κανόνων σε σχέση με το τεκμήριο αθεότητας. Για το τεκμήριο αθεότητα θέλω να πω επίσης ότι η Κομίσιον πήγε πέραν της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υιοθετώντα το δικαίωμα μη αυτοχονοχοποίηση και το δικαίωμα τη σιωπή. Τέλο, η οδηγία η τελευταία οδηγία επιδιώκει έναν βασικό στόχο να εγγυηθεί το γεγονό ότι το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο θα εφαρμόζεται πρακτικά, πράγματι, για τα πιο ευάλωτα άτομα στην αρχή της διαδικασίας, στην πιο κρίσιμη στιγμή για τα άτομα αυτά, τη στιγμή που προφυλακίζονται κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής έρευνας. Η οδηγία λοιπόν σίγουρα δεν περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους κανόνες που προτείνει η Κομισιόν στη συστασή αλλά Ευχαριστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι αν ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε μια οδηγία υιοθετημένη αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βήμα σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Μόνο τέσσερα κράτη-μέλη συμμορφώνονται λίγο πολύ με τις διατάξεις της οδηγίας που έχουμε προτείνει. Θα σταματήσω εδώ. Είχα πολλά άλλα πράγματα να πω βέβαια, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, βρίσκομαι τώρα στη δυσάρεστη θέση να ολοκληρώσω τη σημερινή συζήτηση. Εάν υπάρχει κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση από εσάς, μπορούμε να ε, το κάνουμε ανεπίσημα εδώ μέσα στην αίθουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συμμετέχοντες θερμότατα για τις παρουσιάσεις και τις εισηγήσεις σας. Ευχαριστώ επίσης τους διερμηνείς και ευχαριστώ όλους όσους ήσασταν εδώ σήμερα. Καλό σας βράδυ.